So, nevertheless. Παρά τα αυτά όμως, είναι 3 και 5, ξεκινάμε. Το πρώτο θέμα της ε, σημερινής απογευματινής συνεδρίασης είναι η παρουσίαση του, της Παγκόσμιας Έκθεσης Επενδύσεων του 2017 από την UNCTAD. Με, θέλω να σας παρουσιάσω τον James Chan, ο οποίος προέρχεται από την UNCTAD και είναι διευθυντής του τομέα αυτού. Είναι επίσης και συντάκτης της ετήσιας έκθεσης επενδύσεων. Είναι ο ειδικό για την επενδυτική πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγχαρητήρια στους φιλελεύθερους. Είστε η μεγαλύτερη, πιο πολυάριθμη ομάδα μέσα στην αίθουσα. Η, επενδυτική πολιτική, η πολιτική επενδύσεων εξακολουθεί να είναι ένα από τα ουσιώδη θέματα της ημερήσιας διάταξης. Φυσικά, επίσης, ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών σε περίπτωση επενδύσεων προέκυψε όταν συζητήσαμε την εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία και έχουμε διαφορετικές ε, απόψεις. Η Ιαπωνία λειτουργεί με το παλαιό σύστημα του ISDS και προσπαθούμε τώρα να πείσουμε τους εταίρους μας να περάσουν στο νέο σύστημα το ICTS. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια θετική επενδυτική πολιτική κυρίως από την Κίνα και οι ευρωπαϊκές επενδύσεις ε, στην Κίνα και η πρόταση υπάρχει για το πρασίνισμα των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, όσον αφορά την ψηφιακή πολιτική και τις δυσκολίες ε, λόγω της αλλαγής της βιομηχανικής πολιτικής αποτελούν βασικά θέματα της ε, πολιτικής ξένων επενδύσεων. Υπάρχουν και οι εμπορικές διαστάσεις της ε, ψηφιοποίησης, της ψηφιακής ε, αλλαγής, της ψηφιακής πολιτικής, πολλά ε, καυτά θέματα που έχουν σχέση με τις επενδύσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Τσάν, για να μας δώσετε μια γενικότερη εικόνα του πού βρίσκεται σε παγκόσμιο επίπεδο η πολιτική των επενδύσεων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, ε, ευχαριστώ που καλέσατε την UNCTAD και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ, όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, μετά από πρόσκλησή σας. Θέλω να, εκφράσω και την ευγνωμοσύνη της UNCTAD προς εσάς και τους συνεργάτες σας για την στενή σας συνεργασία με την UNCTAD πέρυσι ε, όπως ιδιαίτερα πέρυσι εσείς συμμετείχατε στο φόρουμ που οργανώθηκε με την ΟΚΤΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα που απασχόλησαν τους πολιτικούς ηγέτες και τους ηγέτες των επιχειρήσεων και που επηρέασε το έργο της ΟΚΤΑΤ. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες. Σήμερα η παρουσίασή μου αφορά τρία θέματα κατά τον α τρόπο ε, θίγονται στην φετινή έκθεση. Πρώτον, είναι οι παγκόσμιες ε, τάσεις στον τομέα των επενδύσεων και οι προοπτικές. Δεύτερον, οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της πολιτικής επενδύσεων, περιλαμβανομένων και κάποια από τα, κάποιων από τα θέματα εθνικής ασφάλειας, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι ενδιαφέρουν τα μέλη εδώ. Και επίσης, ή ε, έχουν σχέση με τη μεταρρύθμιση των επενδυτικών συνθήκων, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε. Και τρίτον, είναι το θέμα της φετινής έκθεσης, είναι η επενδύσεις στην ψηφιακή οικονομία, οι δυσκολίες και οι πολιτικές. Θα ήθελα καταρχήν να σας ενημερώσω για τις ε, ε, παγκόσμιες τάσεις και προοπτικές στον τομέα των επενδύσεων. Το σχεδιάγραμμα δείχνει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι οι τάσεις που θα μπορούσα να πω ε, συνοψίζονται σε χαμηλό επίπεδο ε, ροών επενδύσεων και δύσκολος, δύσκολο δρόμο προς την ανάκαμψη. Δεύτερον, το η γεωγραφική μορφή βλέπουμε ότι οι ροές είναι οι ίδιες ανάλογα με τις περιοχές, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει δραστικά. Κάθε χρόνο αλλάζουν δραματικά. Τέλος, οι προοπτικές. Η UNCTAD είναι ε, έχει μια περιορισμένη αισιοδοξία, περιμένουμε μια μέτρια ανάκαμψη. Και υπάρχει και ένα τελευταίο επιπλέον θέμα που βλέπετε εδώ, όλες αυτές οι επενδυτικές ροές και τάσεις έχουν επιπτώσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες, αξίας και στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ πάλι βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, χρηματοοικονομική κρίση, η επενδύσεις δεν επανήλθαν στο ανώτατο επίπεδο του 2007. Ήδη έχουν μειωθεί κατά 2% σε σχέση με το 34% της αύξησης του 2015. Αν δείτε τα νούμερα θα διαπιστώσετε ότι οι ροές των επενδύσεων βρίσκονται σε ένα δύσκολο δρόμο, δηλαδή έχουν μειωθεί κατά πέντε φορές από την εποχή της κρίσης και ε, μόνο τρεις φορές έχει γίνει προσπάθεια ανάκαμψης. Άρα γι' αυτό λέμε ότι ο δρόμος προς την ανάκαμψη είναι δύσκολος. Δεύτερον, αν δείτε τις επενδυτικές ροές προς ε, ε, περιφέρειες, ας πούμε, τις ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και με, οικονομίες σε μετάβαση, θα δείτε το ίδιο φαινόμενο ότι το 2013 και το 2014 οι ροές επενδύσεως προς τις αναπτυσσόμενες χώρες αυξήθηκαν σημαντικά και ξεπέρασαν τις ε, αναπτυγμένες χώρες συνολικά. Δηλαδή, το μερίδιο των επενδύσεων που πηγαίνει στις αναπτυσσόμενες οικονομίες ήταν μεγαλύτερο από τη ροή των επενδύσεων στις ανεπτυγμένες. Η τάση όμως αυτή αντιστράφηκε το 2015 και το 2016. Τώρα οι αναπτυγμένες χώρες απορροφούν περίπου το 60% των παγκοσμίων ροών των ε, απευθείας ξένων ε, επενδύσεων. Εντός των ανεπτυγμένων χωρών διαπιστώσαμε ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις ε, μειώθηκαν κατά 2%. Ας πούμε, οι ροές επενδύσεων στην Ασία μειώθηκαν κατά 15% και στις περιοχές Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής κατά 14%. Στην Αφρική η μείωση ήταν 5%. Ε, για τις ανεπτυγμένες οικονομίες οι ροές επενδύσεων ήταν σε υψηλό επίπεδο, όμως εξακολουθούν να είναι κατώτερες από το επίπεδο του 1,33 εκατομμύρια δολάρια του 2007. Οι προοπτικές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UNCTAD, οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να μπορεί να αυξηθούν λίγο το 2017 με μια αύξηση περίπου του 5% και να, φτάσουν το 1,753 και να συνεχίσει αυτή η περιορισμένη ανάπτυξη και να φτάσει το 1,853. Κατόπιν αυτού, οι ροές επενδύσεων εξακολουθούν να είναι κατώτερες από το ανώτατο σημείο του 2007. Με, βάση αυτό, αυτή την περιορισμένη αισιοδοξία πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία η οποία θα εμποδίσει τις παγκόσμιες επενδυτικές ροές. πίν το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, το υψηλό επίπεδο πολιτικής αβεβαιότητας και υψηλή γεωπολιτική κίνδυνη και είναι πολλοί και οι άλλοι παράγοντες που θα επηρεάσουν την ανάπτυξη παγκοσμίω των άμεσων ξένων επενδύσεων. Τώρα, οι ροές των παγκοσμίων ε, επενδύσεων και το, οι διάφορες μορφές όπως ας πούμε συγχωνεύσεις και εξαγορές ή εκ του μηδενός επενδύσεις δίνουν κάτι που δεν είναι πολύ ε, καλό για τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες. Αν δούμε τη σύνθεση των ροών των ξένων επενδύσεων παγκοσμίων, αρχικά η όγκος ήταν εξαγορές και ίδιες αναδιαρθρώσεις που συνέβησαν το 2014 και 2015 όταν υπήρξε αύξηση των ε, παγκοσμίων ξένων άμεσων επενδύσεων. Τώρα, οι εκ του ε, οι νέες επενδύσεις δεν έχουν αυξηθεί από την εποχή της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγάλη επέκταση των επιχειρήσεων στις ε, παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Και άρα η, η όθηση του, της, προς την ανάπτυξη του παγκοσμίου εμπορίου, γιατί γνωρίζουμε ότι τα δύο τρίτα του παγκοσμίου εμπορίου πραγματοποιούνται μέσω της, ε, των, παγκοσμίων, της, των παγκοσμίων αλυσίδων αξίας ε, μέσω της διακυβέρνησης. Και ένα τρίτο ε, γίνεται σε εμπόριο στο εσωτερικό των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι ξένες επενδύσεις φέρνουν προηγμένη τεχνολογία, τη γνώση της αγοράς, τεχνογνωσία και δίνουν όθηση στην παραγωγική ικανότητα κυρίως στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπου οι δεξιότητες αυτές και η τεχνολογία ε, λείπουν και χρειάζονται. Και ως εκ τούτου αυτή η τάση ε, εμποδίζει την ανάπτυξη παραγωγικότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Φτάνω τώρα στο δεύτερο σκέλος της έκθεσης, η τις εξελίξεις στον τομέα της επενδυτικής πολιτικής περιλαμβανομένων και των θεμάτων εθνικής ασφάλειας. Θα σας δείξω καταρχήν δύο διαγράμματα που περιγράφουν την δυναμική της πολιτικής αυτής. Υπάρχουν τέσσερα χαρακτηριστικά στις πρόσφατες τέτοιου είδους επενδύσεις, τις ονομάζω τα τέσσερα D. Τη δυναμική στην ε, ε, πολιτική, επενδύσεων, την διχοτόμηση, την διάσταση απόψεων στις ε, ε, ρυθμιστικές τάσεις και την διάσταση στην ε, προσέγγιση προς τις ε, συνθήκες επενδύσεων και το δίλημα στην επιδίωξη των ε, βιώσιμων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Πρώτον, η δυναμική. Τα τελευταίο έτος κυρίως η πολιτική των επενδύσεων υπήρξε πάρα πολύ δυναμική. Πάνω από 50 χώρες έχουν ε, θεσπίσει νέες επενδυτικές πολιτικές με πάνω από 120 μέτρα πολιτικής περιλαμβανομένων και των μεταρρυθμίσεων των εθνικών καθεστώτων ε, επενδύσεων. Μια εξαιρετικά μεγάλη εξέλιξη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αλλά και σε διεθνές επίπεδο συνήφθησαν περισσότερες συνθήκες και είδαμε 30, ε, να συνάπτονται 36 επενδυτικέ συνθήκες και αν συμπεριλάβουμε και αυτές που έγιναν στην αρχή αυτού του έτους είναι άλλες 5. Άρα η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και επιπλέον αν υπολογίσουμε και αυτές που είναι υποδιαπραγμάτευση, διαπιστώνουμε ότι έχουμε πάνω από 100 χώρες να διαπραγματεύονται περισσότερες από 60 συνθήκες τη στιγμή αυτή. Διμερείς, περιφερειακές, υποπεριφερειακές και διαπεριφερειακές. Αυτός είναι ο ρυθμός σύναψης συνθήσεων. Δεν το βλέπουμε σε άλλο χώρο ε, αυτό. Επιπλέον διαπιστώσαμε ότι οι μη ε, δεσμευτικές ε, τάσεις ε, αναπτύσσονται ας πούμε οι νέες ε, ε, πρότυπα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και άλλα. Δηλαδή δημιουργούνται νέα πρότυπα όχι μόνο από κυβερνήσεις αλλά από βιομηχανικές ενώσεις στην κοινωνία των πολιτών ή και από τις ίδιες επιχειρήσεις. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που ανέφερα είναι η διάσταση απόψη, η διχοτόμηση των κατευθύνσεων, των ρυθμιστικών κατευθύνσεων. Αριστερά στο διάγραμμα βλέπετε ότι σε εθνικό επίπεδο η πολιτική ε, προχωρεί παράλληλα. Δηλαδή βλέπουμε ταυτόχρονα απελευθέρωση, προώθηση των επενδυτικών μέτρων μαζί με την αύξηση των περιορισμών και των προστατευτικών μέτρων απέναντι στις επενδύσεις βλέπουμε ότι καμιά φορά και οι ίδιες χώρες θεσπίζουν μέτρα και απελευθέρωσης και πρόθεσης και μέτρα περιορισμού και προστατευτισμού ταυτόχρονα. Αυτό ονομάζω εγώ διχοτόμηση, διάσταση. Αν δείτε το αριστερό σκέλος στις αρχές της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του αιώνα μας βλέπετε ότι κατά μέσο όρο 9% των νέων μέτρων που θεσπίζονταν από τις χώρες πήγαιναν προς την κατεύθυνση του περιορισμού. Τώρα 30% των μέτρων είναι περιοριστικά και προστατευτικά συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων εθνικής ασφάλειας επί των οποίων θα επεκταθώ αργότερα. Στο δεξί μέρος της εικόνας βλέπετε τη δυναμική της ε, δια, διεθνούς τάσης σύναψης θε, ε, συνθήκων και το, ονομάζω ε, διάσταση γιατί αυτή τη στιγμή ασκούνται τέσσερις δυνάμεις υπάρχουν χώρες ε, που συνάπτουν νέες συνθήκες, στις οποίες προσπαθούν να αυξήσουν τη συνθή, την προστασία των επενδύσεων και να συμπεριλάβουν ε, τις διαστάσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό το ονομάζουμε άνοδο ε, και ενημέρωση των του επίπεδου των διεθνών συνθήκων. Και υπάρχουν και οι χώρες, απ' την άλλη, που απεμπλέκονται από τα διάφορα, από το καθεστώς διεθνών επενδύσεων, απομακρύνονται από τις συνθήκες, φεύγουν από το σύστημα και αποδεσμεύονται από τις πολυμερείς διαδικασίες. Ε, αυτή είναι η δεύτερη δύναμη κάποιες χώρες πραγματικά ε, σταματούν την συμμετοχή τους. Πέρυσι έληξαν 19 συνθήκες, μάλλον 19 συνθήκες, από 19 συνθήκες αποχώρησαν χώρες. Και υπάρχουν ε, κάποιες ε, που είναι βασικές δυνάμεις αναδιόμενες. Κατόπιν υπάρχουν χώρες που αναθεωρούν και ανα... αλλάζουν τα μοντέλα συνθήκων, τις διαπραγματευτικές τους θέσεις και ετοιμάζονται να διαπραγματευτούν ε, επενδυτικές συνθήκες νέας γενιάς. Αυτό έχει σχέση με αυτό που ονομάζω εγώ την μεταρρύθμιση των ε, καθεστώτων διεθνών επενδυτικών συνθήκων. Ο πρόεδρος πριν από λίγο αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της UNCTAD για τη μεταρρύθμιση των ε, εθνικών επενδυτικών ε, καθεστώτων του 2013, εμείς χωρίσαμε τις φάσεις της μεταρρύθμισης σε δύο τη μεταρρυθμίσει σε δύο φάσει. Η πρώτη προχωρεί πάρα πολύ καλά και έχουν επιτευχθεί σπουδαία πράγματα. Τι εννοούμε πρώτη φάση. Είναι η φάση κατά την οποία οι χώρε ή οι περιφερειακές ε, ομάδες χωρών αναθεωρούν ε, τις συνθήκες τους, αναθεωρούν τις θέσεις τους και ετοιμάζονται για διαπραγματεύσεις. Το γεγονός ότι αυτή η νέα γενιά ε, μοντέλων επενδυτικών συνθήκων ε, οδηγεί στη διαπραγμάτευση νέων συνθήκων. Αυτό έχει συμβεί. Το βλέπουμε. Και η έρευνα ε, στις ε, νέα, ε, συνθήκες νέας γενιάς που υπογράφηκαν τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια μας δείχνουν ότι υπάρχει η τάση να ενταχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στο σώμα των συνθήκων με μια εξισορρόπηση ε, μεταξύ των κρατών και των επιχειρήσεων. Αυτή είναι μια θετική τάση. Η δεύτερη φάση μεταρρύθμισης θα αφορά τις ε, υπάρχουσες, τις υφιστάμενες συνθήκες πάνω από 2.700 επενδυτικές συνθήκες παλαιάς γενεάς όπως τους ονομάζουμε που έχουν συναυθεί στις δεκαετίες του 80, του 90 και στις αρχές του 21ου αιώνα πριν τη χρηματοοικονομική κρίση, πριν την αλλαγή του προτύπου προς τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι συνθήκες αυτές είναι πολλές και δύσκολες και αν δείτε τις περιπτώσεις διευθέτησης διαφορών τα τελευταία χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι όλες αυτές οι περιπτώσεις, προκύπτουν από τις παλαιάς γενεάς συνθήκες και βλέπουμε ότι πάνω από το 95% των συνθήκων δεν αναφέρουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν έχουν μια διάσταση βιώσιμης ανάπτυξης, δεν προβλέπουν τη ρύθμιση στοιχείων τέτοιου είδους. Οπότε πρέπει να ασχοληθούμε με τις συνθήκες αυτές. Αυτή είναι η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης. Και στην έκθεση φέτος αναφέρουμε δέκα δυνατότητες αντιμετώπισης των συνθήκων αυτών παλαιάς γενεάς. Εξυγχρονισμό, ενημέρωση ή και χρήση διαφόρων μέτρων ώστε να τις αναβαθμίσουμε για την αποφυγή των διαφωνιών που θα εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της διάστασης ε, των προσπαθειών για τη σύναψη συνθήκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως, στο τομέα των διεθνών επενδυτικών πολιτικών είναι, υπάρχει αυτό που ονομάζω δίλημα. Ποιο είναι το δίλημα. Σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον οι ηγέτες, οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες έχουν δεσμευτεί στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε θεσπίσει 17 ε, στόχους και οι χώρες ε, υιοθετούν πολιτικές. Όλοι οι περισσότεροι από αυτούς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης αφορούν κλάδους της ε, βιομηχανίας που είναι πολύ ευαίσθητοι για τις κυβερνήσεις γεωργία, υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες όπως παροχή ύδατος, αστική ανάπτυξη και άλλα τέτοια θέματα. Και αυτοί είναι τομείς που χρειάζονται σαφώς επενδύσεις και υπάρχει ένα χρηματοδοτικό χάσμα 2,33 ευρώ ε, δολάρια το χρόνο για κάθε κλάδο. Χρειάζονται λοιπόν ε, ιδιωτικές επενδύσεις σε αυτούς τους χώρους. Όμως, στους χώρους αυτούς, αν δείτε τις επενδυτικές πολιτικές, διαπιστώνετε ότι είναι η περισσότερο κλειστή σε ξένες ή ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό είναι ευνόητο φυσικά, είναι κατανοητό, διότι εκεί χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις, ούτω ώστε να παρέχονται αγαθά και υπηρεσίες σε με τρόπο που να είναι προσβάσιμο και για στους φτωχούς και να έχουν τη δυνατότητα να τις πληρώσουν οι φτωχοί. Αυτό όμω είναι δύσκολο και αυτό ακριβώς είναι το δίλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτοί που θεσπίζουν την πολιτική και οι νομοθέτες όπως εσείς. Υπάρχει η ανάγκη εξισορρόπησης των ιδιωτικών με τις δημόσιες επενδύσεις, να εξισορροπηθούν οι ανάγκες, να βελτιωθούν οι κίνδυνοι και το αποδοτικό προφίλ των επενδύσεων και η ανάγκη να εξασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, οι δημόσιες υπηρεσίες, ότι θα παρέχονται σε, σε κατάλληλο κόστος ε, υπηρεσίες στους φτωχούς για να έλθω τώρα σε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ, το θέμα της εθνικής ασφάλειας. Αν δείτε τα γραφήματα, στο πρώτο βλέπετε ότι οι εξαιρέσεις της εθνικής ασφάλειας που έχουν ε, θεσπιστεί στις ε, διεθνείς ε, συμβάσεις έχουμε μια βάση δεδομένων με χιλιάδες επενδυτικές συνθήκες και έχουμε παρακολουθήσει αυτές τις συνθήκες για να δούμε πώς οι εξαιρέσεις της εθνικής ασφάλειας αντικατοπτρίζονται στις συνθήκες αυτές ε, μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Αν δείτε εδώ, βλέπετε ότι βασικά Καταρχήν, η κάλυψη όλων των επενδυτικών ε, συνθήκων ε, φαίνεται να είναι πολύ χαμηλή και αν δείτε τις συνθήκες που υπογράφησαν μέχρι το 2000, είχαμε μόνο 9% των συνθήκων που κάλυπταν ε, αυτές τις εξαιρέσεις εθνικής ασφάλειας. Και συνολικά, με όλες ε, τις ε, συνθήκες, βασικά μόνο το 14% καλύπτουν θέματα εθνικής ασφάλειας και μιλάμε περίπου για 350 τέτοιες συνθήκες. Όμως, αν δείτε τις πιο πρόσφατες που υπογράφησαν μεταξύ του 2011 και του 2016, το ίμιση αυτών καλύπτουν εξαιρέσεις εθνικής ασφάλειας. Αυτό μας δείχνει ότι δίνεται μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα εθνικής ασφάλειας ε, κατά τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε την ε, επισκόπηση της ε, στρατηγικής εθνικής ασφάλισης και κάναμε μία έρευνα όλων περιπτώσεων, πάνω από 50 χώρες, μεγάλες οικονομίες, εδώ μιλάμε για μεγάλες οικονομίες, έτσι λοιπόν, πάνω από 50 χώρε ε, έχουν περιορισμού επενδύσει σε ευαίσθητου τομεί, 14 χώρε ε, έχουν κρατικά μονοπόλια και ξεκάθαρη νομοθεσία. Και ουσιαστικά μιλάμε ότι επιτελούν δραστηριότητες για βασικές δημόσιες υπηρεσίες και έχουμε κάποιες άλλες χώρες με μηχανισμούς αναθεώρησης για προκαθορισμένους τομείς που απελευθερώνουν αλλά θέλουν να παρακολουθούν και κατόπιν έχουμε 8 χώρες ε, με ε, μηχανισμούς ελέγχου για τις ξένες επενδύσεις, ε, δηλαδή απελευθερώνουν, δεν περιορίζουν τους τομείς, αλλά έχουν ουσιαστικά θεσπίσει ένα μηχανισμό παρακολούθησης. Επίσης, βλέπουμε νέα μέτρα πολιτικής που έχουν θεσπιστεί μεταξύ του 2006 και του 2016, τα τελευταία δεκαέτη. 22% των, πολιτικών, των νέων πολιτικών σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια. Και αυτό σχετίζεται με την αναθεώρηση των εθνικών στρατηγικών, με τους μηχανισμούς αναθεώρησης, ε, με διάφορες διαδικασίες που σχετίζονται με τον έλεγχο της εθνικής ασφάλειας. Τώρα, ποια άλλα θέματα πολιτικής εμπλέκονται σε αυτό τον έλεγχο εθνικής ασφάλειας. Έχουμε τέσσερα κυρία θέματα μεταξύ άλλων. Καταρχήν, οι χώρες έχουν διάφορα είδη κανονισμών άμεσων ξενών επενδύσεων ε, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Δεύτερον, οι διαδικασίες ελέγχου των επενδύσεων χρησιμοποιούν ε, διάφορες ενίες ε, για την εθνική ασφάλεια. Τρίτον, οι χώρες διαφέρουν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και το βάθος των διαδικασιών ελέγχου των επενδύσεων. Και τέταρτον, πολύ σημαντικό, είναι το πώ ε, να διαχωρίσεις τι νόμιμες ανησυχίε της κοινή γνώμη έναντι των προστατευτικών μέτρων. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και λέμε ότι ο προστατευτισμός ε, ε, ουσιαστικά εξαρτάται από αυτόν που τον ασκεί, γιατί δεν υπάρχει ορισμός ε, του προστατευτισμού στο στάδιο αυτό σε κανένα μέσο διεθνούς πολιτικής. Τώρα έρχομαι στο τελευταίο μέρος το οποίο σχετίζεται με το θέμα της φετινής έκθεσης, επενδύσεις ε, στην ψηφιακή οικονομία, πολιτικές και προκλήσεις. Εδώ στο γράφημα βλέπετε τους κύριους πρωταγωνιστές ε, των παγκοσμίων αλυσίδων αξία, των ψηφιοποιημένων αλυσίδων αξία. Ε, νομίζω ότι πλήττονται πάρα πολύ από την ψηφιοποίηση, θίγονται πάρα πολύ από την ψηφιοποίηση της οικονομίας παγκοσμίω, επομένως ε, θα έχουν αντίκτυπο στο εμπόριο και στις επενδύσεις. Για να το τονίσω, καταρχήν, η ψηφιοποίηση μεταμορφώνει την ε, διεθνή παραγωγή και τις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής. Ο αντίκτυπος τη ψηφιοποίηση στην ε, διεθνή παραγωγή εμπλέκει όλους τους παράγοντες των ψηφιακών οικοσυστημάτων. Εδώ αναφέρουμε τεχνολογίες πληροφοριών και τεχνολογιών, ε, τις πολυεθνικές, τις ψηφιακές πολυεθνικές και τις παραδοσιακές πολυεθνικές. Πώς ε, αυτά θίγουν ε, τις εταιρείες και τις συναλλαγές τους παγκοσμίω, το ουσιαστικά μεταμορφώνουν το παγκόσμιο τοπίο. Καταρχήν έχουμε νέους παίκτες, όπως είναι οι τεχνολογίες πληροφοριών, και δρούν ε, πάρα πολύ ε, γρήγορα, γρηγορότερα από τις παραδοσιακές πολυεθνικές. Αν δείτε την κατάταξη των ε, πρώτων 100 ή 500 πολυεθνικών βλέπουμε όλο ένα και πιο ψηφιακές πολυεθνικές να κινούνται πιο πάνω στην κατάταξη, πολύ ταχύτερα από άλλες εταιρείες. Δεύτερον, πρώτη φορά η Εκτότη κάνει έναν κατάλογο των 100 ε, ε, μεγαλύτερων πολυεθνικών ε, και βλέπουμε ότι όσε είναι ψηφιακέ αναπτύσσονται πολύ γρηγορότερα. Ουσιαστικά διαφέρουν αυτές οι πολυεθνικέ από τις παραδοσιακέ. και αν δείτε το διεθνέ αποτύπωμά τους έχουμε τρία κυρία χαρακτηριστικά. Καταρχήν, έχουν ένα ε, ελαφρό έχουν ελαφρά διεθνή περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή λιγότερες ξένες επενδύσεις. Ε, δεύτερον, έχουν υψηλή συγκέντρωση. το σχάρι. αν δείτε τις ε, κορυφαίες εταιρείες, το 60% με, από αυτές τις εταιρείες έχουν έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα άλλο ένα 30%. Είναι τοποθετημένε μόνο σε λίγε χώρε όπω στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Κορέα και τη Γερμανία. Πολύ λίγε. Έτσι λοιπόν, ε, έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση από τι παραδοσιακέ πολυεθνικέ και αυτό φυσικά έχει συνέπειε στον ανταγωνισμό. Υπάρχουν θέματα παγκόσμιου ανταγωνισμού. Τρίτον, έχουν ε, ε, ουσιαστικά μεγάλα χαρτοφυλάκια απολύσεων και μετρητών στο εξωτερικό και αυτό φυσικά έχει συνέπειες στα φορολογικά εισοδήματα των χωρών. Αυτά είναι τα κύρια τρία χαρακτηριστικά που μπορείτε να θέλετε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, η ψηφιοποίηση των οικονομιών επίσης ε, θίγει τις παραδοσιακές πολυεθνικές εταιρείες ε, με σημαντικό τρόπο και θα σας παρουσιάσω τρία χαρακτηριστικά. Καταρχήν, η ψηφιοποίηση φύγει οποιοδήποτε τμήμα ολόκληρων των αλυσίδων αξίας, ε, είτε μιλάμε ε, για την παραγωγή, την έρευνα και την ανάπτυξη, ε, την επιμελητία, τις σχέσεις με τους πελάτες και την δομή της διακυβέρνησης της πολυεθνικής, της πολυεθνικής ακόμη και τις δημόσιες συμβάσεις. Δεύτερον, υπάρχει μία μετάβαση προς ε, ένα, μια, ένα αφρύτερο τρόπο πραγωγής. Τι εννοώ, το ανέφερα αυτό νωρίτερα. Δηλαδή, θα υπάρχουν ολένα και λιγότεροι τρόποι επένδυσης σε ίδια κεφάλαια, σε άμεσες εξένες επενδύσεις. Ουσιαστικά, χρησιμοποιούν περισσότερο ε, τρόπους όπως είναι η αδειοδότηση, το franchising, διάφορες συμβάσεις. Έχουμε δύο λόγους για τη μετατροπή των κινδύνων, επειδή υπάρχουν διάφορες αβεβαιότητες σήμερα και λόγω και της ε, ψηφιοποίησης. Τρίτον, έχουμε αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα, αντιδοκοποιούν τις διεθνείς ε, συναλλαγές τους ε, και ουσιαστικά ε, διαλύουν τα επιχειρηματικά μοντέλα των παραδοσιακών πολυεθνικών. Παραδείγματο χάρη έχουμε διάφορα μοντέλα ε, όπως υπάρχει η μη διαμεσολάβηση, διευρυμένη μεσολάβηση, η ευέλικτη παραγωγή, η διανεμημένη παραγωγή. Έχουμε λοιπόν διάφορα τέτοια νέα μοντέλα επιχειρηματικά. Αυτό είναι ο αντίκτυπο. Το δεύτερο μήνυμα κλειδί που θέλω να στείλω μέσω της έκθεσης είναι ότι είναι εφικτό το ίντερνετ, το διαδίκτυο για όλους. Το βλέπουμε αυτό στο άμεσο μέλλον. Τι σημαίνει αυτό. Στους στόχους της ε, χιλιετίας ε, έχουμε το στόχο να υπάρχει παγκόσμια σύνδεση στο ίντερνετ και νομίζουμε ότι είναι ε, εφικτό. Υπολογίσαμε ποιο είναι το ψηφιακό χάσμα για να υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ, διαθεσιμότητα στο ίντερνετ για όλους και υπολογίσαμε τι χρειαζόμαστε. Αν ε, θέλουμε να καλύψουμε αυτό το κενό της, της συνδεσιμότητας στο ίντερνετ, τουλάχιστον σε κάλυψη ευρυζωνική 3G για διάφορες χώρες ε, και οικονομία σε μετάβαση. Δεν θέλουμε πολλές επενδύσεις. 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα αρκούσαν για να φτιάξουμε την βασική συνδεσιμότητα σύνδεση στο ίντερνετ 3G ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις μεταβατικές οικονομίες. Λεχθέντως αυτού, Χρειαζόμαστε και άλλες ε, πτυχέ που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, δηλαδή τη συνδεσιμότητα των επενδύσεων θα πρέπει να υποστηρίζεται από υποδομή ε, ηλεκτροδότησης στις στοχότερες χώρες. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε και ανάπτυξη δεξιοτήτων, παροχή περιεχομένου και διαθεσιμότητα προκειμένου να μειωθεί το κενό της υιοθέτηση. Έχουμε δηλαδή την ευρυζωνική κάλυψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί ο πληθυσμό να έχει πραγματική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έτσι, λοιπόν, χρειαζόμαστε διαθεσιμότητα. Νομίζω ότι καθυστέρησα πάρα πολύ, φτάνω προς το τέλος. Ερχόμαστε με ένα πλαίσιο πολιτικές για την επένδυση στην ψηφιακή οικονομία. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση το πλαίσιο, καταρχήν ξεκινάμε τις στρατηγικές για την ανάπτυξη των ψηφιακών οικονομιών, κυρίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες, υπό το φως της συγκέντρωσης των ψηφιακών εταιριών. Στην περίπτωση αυτή, θέλουμε να εντάξουμε τις επενδυτικές πολιτικές ε, στις στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και αντιστρόφως. Μέχρι τώρα, βλέπουμε έλλειψη και στα δύο. Και σε ψηφιακές οικονομίες η ανάπτυξη σημαίνει όχι μόνο την ανάπτυξη υποδομής, αλλά και των ψηφιακών εταιριών, του ψηφιακού τομέα, αλλά και την οθέτηση της ψηφιοποίησης σε όλους τους τομείς. Ιδίω για τις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να μπορέσουν ε, να ακολουθήσουν τις εξελίξεις ε, και να είναι ανταγωνιστικές ε, στις διεθνείς αγορές για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Και βεβαίως θα πρέπει να εξισορροπήσουμε το δημόσιο συμφέρον με το ιδιωτικό συμφέρον, γιατί ξέρουμε ότι θα πρέπει να εξαλείψουμε τα εμπόδια για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Και αυτά τα εμπόδια επίσης μας δείχνουν τις ανησυχίες ε, δημόσιου χαρακτήρα. Πρέπει λοιπόν να τα ξεσορροπήσουμε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ε, πολύ ενδελεχή ματιά παγκοσμίω. Λοιπόν, τώρα θα δώσω το λόγο σε εσά, αγαπητοί συνάδελφοι. είναι πρώτα και υπόλοιποι εργότερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας που μας έδωσε ουσιαστικά μια ευρύ εικόνα για τις άμεσες ξένες επενδύσεις ε, στις αλυσίδες αξίας. Θέλω να σας θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι προφανές ότι για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε πολλές επενδύσεις στις χώρες όπου απαιτείται αυτό περισσότερο, όπου απαιτούνται και οι απαραίτητε υποδομές, χρειάζεται μία συνεργασία δημοσιοδιωτικού τομέα. Όμως, επίσης, πρέπει στις χώρες αυτές οι κυβερνήσεις να έχουν το κατάλληλο προσωπικό για να μπορεί να ελέγξει και να παρακολουθήσει αυτούς τους επενδυτικούς μηχανισμούς. Πολύ συχνά βλέπουμε ότι τα κέρδη είναι ιδιωτικά, αλλά οι απώλειες είναι δημόσιες, γιατί υπάρχουν λάθη στο μοντέλο, στην εφαρμογή, στον έλεγχο και τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά. Και αυτό οδηγεί στο να έχει αρνητική εικόνα ο μηχανισμός. Από την άλλη υπάρχει ένα θέμα που δεν θύχτηκε. Δύο θέματα. Θα ήθελα τη γνώμη σας γι' αυτά. Καταρχήν, εγώ νομίζω ότι σχετίζεται πάρα πολύ το θέμα της προσέγγισης επενδύσεων, ε, το θέμα των φορολογικών εκτόσεων, Δηλαδή, κάποιες ε, χώρες ε, προσφέρουν φορολογικά κίνητρα και εκπτώσεις για να ε, σταματούν οι εταιρείε να πληρώνουν φόρους, όμως αυτό δεν είναι κάτι θετικό. Εσείς εργάζεστε ουσιαστικά προς κάποια νομοθεσία έτσι ώστε να υπάρχει μια φορολογική διακυβέρνηση και να πληρώνουν οι επιχειρήσεις για τα κέρδη τους και να σταματήσουν τα κράτη να ελκύουν επενδύσεις επειδή δεν πληρώνουν οι εταιρείε φόρους. Επίσης, για το δημόσιο σύστημα επενδύσεων, στο οποίο εργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει συμπεριληφθεί στη συμφωνία με τον Καναδά και το οποίο τελικός στόχος είναι να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πώς βλέπετε το σχεδιασμό αυτού του μαντέλου και ποιες ε, δυνατότητες βλέπετε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολυμερώς. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σάκη, ευχαριστώ πολύ. Δεν σα άκουσα στην αρχή, την περιμένω να τελειώσει η διερμηνία στη γλώσσα μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαν για την εξαιρετική σας παρουσίαση. Ήταν πάρα πολύ επίκαιρη κιόλα. Ασχολήθηκε με όλα αυτά τα καυτά πολιτικά ζητήματα που αφορούν και εμάς. Είμαι συντάκτρια τη έκθεση για το ψηφιακό εμπόριο. Έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και στο παρελθόν και συμφωνώ ότι υπάρχουν ταχύτατε εξελίξει στον κλάδο και πρέπει να προσπαθήσουμε να τι καταλάβουμε και τι ενώσουμε. Καταλαβαίνω όμω ότι και αυτή η συζήτηση είναι αρκετά πολιτική και προ τα εκεί θα κινηθούν οι ερωτήσει μου. Έτσι ώστε να προσπαθήσω να ρίξω μια πιο προσεκτική ματιά στι συνέπειε αυτού που κάνουμε τώρα. Κάτι που φάνηκε στην παρουσίασή σας είναι η ανάγκη για άμεσες επενδύσεις και για να καταλάβουμε επίσης πως υπάρχουν και στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. Ταυτόχρονα όλες οι συνθήκες, οι ε, μακροχρόνιες συνθήκες που έχουν και προστασία των επενδυτών πρέπει να ελέγχονται επαρκώς. Ε, ιδιαίτερα εκείνοι που πιστεύουν στην ανάπτυξη πρέπει να ασκήσουν και μεγαλύτερο έλεγχο στις παλαιότερες συνθήκες. Επίσης υπάρχει ένας κίνδυνος για να... Υπάρχει και ένας κίνδυνος να μην προχωρήσουμε όταν ε, φοβούνται να επαναεξετάσουν και να αναθεωρήσουν τις συνθήκες ή να μην συμπεριλάβουν όλες τις ε, διατάξεις που πρέπει, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη συμφωνία με την Ιαπωνία. Επίσης, ε, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον ότι όσο πιο συντηρητικός είναι κάποιος, ε, τόσο, πιο, ε, τόσο περισσότερες εξαιρέσεις ε, ζητά σε συμφωνίες για άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη. Και αυτό μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Να σας ρωτήσω επίσης για τον κίνδυνο παράλυσης, για τον κίνδυνο στασιμότητας στους κανόνες και εσείς ε, τι πιστεύετε πως αυτό θα επιφέρει στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και στις επενδύσεις της ίδιες. Και μετά, ε, η σημασία του διαδικτύου για όλους, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Εσείς πώς βλέπετε το ρόλο του ιδιωτικού τομέα απέναντι στον δημόσιο και αναφερθήκατε σε ορισμένες επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ισορροπία ανάμεσα στις πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες που έχουν και την εξουσία για να λαμβάνουν αποφάσεις και στις ε, μικρότερες. Εκεί υπάρχει άμεση σχέση με τις α, ξένες επενδύσεις. είναι οι επιπτώσεις και ποια είναι τα ωφέλη του διαδικτύου για όλους που παρέχεται από δημόσιους φορείς με εκείνους που παρέχονται από, από ιδιώτες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, θα ήθελα να μάθω και για το πώς συνδέονται αυτοί οι τομείς, ποια είναι η διάδραση μεταξύ τους στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπου μπορεί να επικρατήσουν επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ. Ο Χέλμου Τσόλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζάν για την πολύ λεπτομερή παρουσίαση, τα ευρήματα του 2017 αφού είχαμε την ανταλλαγή απόψεων νωρίτερα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω να, τα, να ακούσουμε αυτά που είχατε να μας πείτε. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για τις επενδυτικές πολιτικές που έγιναν στους διάφορους τομείς που μας αναφέρατε. Αυτές οι πολιτικές έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη, στη βιομηχανία, στις υποδομές, όπου αυτές εφαρμόστηκαν. δεν αναφέρομαι τόσο στις αξίες, στην αξία των επενδύσεων, αλλά ποια ήταν η ποιότητα. Έφεραν αυτές, αυτή τη διαφορά, έκαναν κάτι το οποίο είχε μακροπρόθεσμες ε, επιπτώσεις και μακροπρόθεσμα ωφέλη, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας δείξετε με κάποια παραδείγματα πώς οι διασυνοριακές επενδύσεις, είτε αυτές είναι ιδιωτικές είτε αυτές είναι δημόσιες, έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη αυτή. Και οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτές τις επενδυτικές πολιτικές συμμορφώνονται με τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει μήπως ανάγκη να κάνουμε περισσότερα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ζαν για την εξαιρετική του παρουσίαση σχετικά με τις επενδύσεις. Όπως είπε και ο κύριος Σόλτς μόλις τώρα, η ποιότητα των επενδύσεων είναι σημαντική. Και η πρώτη μου ερώτηση αφορά αυτό. Μας είπατε ξεκάθαρα ότι το επενδυτικό κενό που υπάρχει είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί έτσι ώστε να ε, τηρήσουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και τους στόχους της χιλιετίας. Είναι τεράστιο αυτό το κενό. Αλλά ας δούμε τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το σκεπτικό πίσω από αυτό ήταν να καλέσουμε τον ιδιωτικό τομέα να ε, συνεισφέρει στους ε, στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης μέσω οικονομικών κινήτρων δημοσίου. Αυτό είναι κάτι που συζητά πολύ καιρό το Κοινοβούλιο και το κατάφερε, το δημιούργησε μετά από πολύ αγώνα. Εσείς πώς νομίζετε πώς μπορεί να συνεισφέρει και ποιοτικά, όχι μόνο ποσοτικά. Μετά, οι προποθέσει για τις επενδύσεις. Πολλές φορές υπάρχουν αυστηρά κριτήρια. Υπάρχει αυστηρότατος και τεράστιος ανταγωνισμό ανάμεσα σε χώρες. Η UNCTAD τι κάνει γι' αυτό, πώς ε, διαδραματίσει συμβουλευτικό ρόλο, τι κάνει για να αποφύγουν ε, την φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή, την κλεπτοκρατία, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και τρίτη ερώτηση, τι νομίζετε και ποια είναι η άποψή σα για την πρωτοβουλία της κυρίας Μάλιμστρομ για το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο. Θεωρείτε πως οι δασμοί για τις επενδύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον δημιουργηθεί τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ. Με το λόγο βάσει ενός εγγραφού που μου ζήτησε ο κύριος Μουλής σας Έχει τέσσερις ερωτήσεις να θέσει για την ε, έκθεση. Το πρώτο, κατά την έκθεση ανάγνωση της έκθεσης του 2017 για τις παγκοσμίες ε, επενδύσεις του φαίνεται ότι υπάρχει ένα διπλό φαινόμενο που μπορεί να φαίνεται παράδοξο. Καταρχήν ε, υπάρχει μία σειρά έκρηξης μέτρων απελευθέρωσης των επενδύσεων ε, και το ίδιο έτος μείωση του ποσοστού των διεθνών επενδύσεων με αρκετά μετριοπαθείς δυνατότητες προοπτικές ανάπτυξης. Υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ ε, του πολλαπλασιαστή της πρόθεσης των επενδύσεων και του πραγματικής ροής των επενδύσεων αυτών. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το καθεστώς προστασίας των επενδύσεων Υπογραμμίζει η έκθεση ότι ε, πολλές διαδικασίες επίλυσης ε, διαφορών τύπου SDS παραμένουν ε, πολύ υψηλές και 60% κερδίζουν οι επενδυτές και είπατε ότι έγινε πρόοδος ε, ως προς τη μεταρρύθμιση ε, των μηχανισμών προστασίας των επενδύσεων βάσει του κεφαλαίου της προστασίας των επενδύσεων που έχουμε τώρα στη ΣΕΤΑ και αναμένοντας ε, ένα, τη δημιουργία ενός διαφορετικού συστήματος επίλυση διαφορών, τι θα συστήνατε εσείς. Επίσης, έχουμε συγκεκριμένο θέμα για την εφρική η Αφρικανική βλέπει ένα έλλειμμα επενδύσεων, μείωση 3% για το 2016. Αν ε, βλέπει η Αφρική μία μείωση, ε, βλέπει και μείωση υπεύθυνων επενδύσεων ως προς σεβασμό ε, του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα μέσο όπως το σχέδιο Juncker για την άφηση μπορεί να δώσει όθηση στις επενδύσεις για την Αφρική και πώς ε, ε θεωρείτε ότι θα υπάρχει πραγματική ανάληψη ευθύνη από τις πολυεθνικές για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με πιο τομεακή πτυχή ε, πρόσφατα τέθηκε το θέμα του ελέγχου των επενδύσεων στους στρατηγικούς ε, τομείς ε, στα θεσμικά όργανα. Έχουμε ε, κατά νου κάποιες επενδύσεις επιθετικές όπως της Κίνας στην Ευρώπη. Αυτή η τάση επενδύσεων παρατηρείται σε στρατηγικούς τομείς και ναι, βλέπετε να υπάρχει επιτάχυνση αυτού του φαινομένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και εγώ δύο ερωτήσει για εσά, κύριε Ζαν. Η μία αφορά το πρασίνισμα των επενδύσεων. όπου υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι ένα υπαρκτό μέσο, είναι πραγματικό ή είναι πιο πολύ κάτι που χρησιμοποιούμε για να δείξουμε πολιτική ισχύ. Και Πόσο συχνά χρησιμοποιούμε κάτι τέτοιο ή μήπω είναι κάτι που χρησιμοποιούμε έτσι αποτρεπτικά. Μετά, η δεύτερη μου ερώτηση μοιάζει με αυτή που έκανε η συνάδελφος πιο πριν. Η συγκέντρωση των επενδύσεων στον ψηφιακό κόσμο. Εάν θέλουμε να προωθήσουμε επενδύσεις και αν προωθούμε την ψηφιοποίηση, πώς μπορούμε να αποφύγουμε ότι αυτή η τάση συγκέντρωση των επενδύσεων σε συγκεκριμένες εταιρείες, ελάχιστες εταιρείες, κυρίως εταιρείες οι οποίες βρίσκονται εκτός από τις χώρες τις οποίες στοχεύουμε να επενδύσουμε, πώς ε, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τις ε, συνθήκες έτσι ώστε να αποφεύγουμε κάτι τέτοιο. Πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια τέτοια συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείξατε για αυτό που κάνουμε στην UNCTAD και βλέπω πως οι αγαπητοί ευρωβουλευτές έχουν διαβάσει πολύ προσεκτικά την έκθεση για τις παγκόσμιες επενδύσεις. Τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει ότι στις επαφές μου μαζί σας οι ερωτήσεις σας γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες και ολοένα και περισσότερο επί της ουσίας. Μου κάνετε λοιπόν πιο δύσκολη τη ζωή. Σας ευχαριστώ πρώτη ερώτηση που αφορούσε την ανάγκη για επενδύσεις σε επιχειρήσεις, την ανάγκη δημιουργίας ικανοτήτων για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πράγματι, δημιουργούμε ικανότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες, έτσι ώστε να τις βοηθήσουμε να δημιουργήσουν μια νέα γενιά επενδυτικών πολιτικών. Έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής ε, στον οργανισμό μας και τον χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να αναθεωρήσουν τις επενδυτικές τους πολιτικές. Ιδιαίτερα οι κυβερνήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν ε, για πρώτη φορά την εξουσία. Επίσης προσπαθούμε να καταρτήσουμε προσωπικό, να καταρτήσουμε τους ε, διαπραγματευτές, λειτουργούμε συμβουλευτικά και όπως είπατε και εσείς, αυτό το έργο μας είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια νέα γενιά επενδυτικών πολιτικών που θα συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε το, τη σύνδεση των φορολογικών κινήτρων και ε, ωφελιών στις, ε, για να δημιουργηθούν και να γίνουν ξανά επενδύσεις. θεωρούσαμε στο παρελθόν ότι οι επενδύσεις που θα προσελκύσουν επενδύσεις είναι λίγο το κεραστάκι στην τούρτα, γιατί οι επενδυτές αυτό που ψάχνουν είναι να βρουν, για παράδειγμα, στοιχεία όπως το μέγεθος της αγοράς, την πολιτική, τη διαφάνεια, σταθερότητα μιας αγοράς, υποδομές, εγκαταστάσεις κτλ. Υπάρχουν λοιπόν τρεις ε, ομάδες καθοριστικών παραγόντων η... τα κίνητρα για τους επενδυτές είναι το κερασάκι στην τούρκετα. Είναι αυτό που θα εξετάσουν αφού εξετάσουν όλα τα προηγούμενα. Όμως, τούτου λεχθέντος να πω ότι για τις φτωχότερες χώρες με τα χαμηλότερα εισοδήματα, ο κίνδυνος ε, για να αποβεί κερδοφόρα μια, επιχει... μια επένδυση είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους επενδυτές. Πολλές φορές λειτουργεί αποτρεπτικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εκεί είναι να δημιουργήσουμε ε, επενδύσεις οι οποίες ε, θα ε, δημιουργήσουν πιο προσβα... συνθήκες πιο προσβάσιμες για τους πολίτες, για τους φτωχότερους πολίτες. Όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος και δεν είναι ελκυστική μια επένδυση, τότε χρειαζόμαστε πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική για να έχουμε απόδοση αυτή τη επένδυση σε βάθο χρόνου και ίσω οι επενδυτές ε, το χρειάζονται κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να έχουν αυτή την ε, σιγουριά σε βάθο χρόνου και όταν είναι δύσκολο για χώρα να δώσει αυτά τα κίνητρα στους επενδυτές, εμείς ε, παίζουμε ένα ρόλο. Εμείς κοιτάμε τα παραδείγματα στο παρελθόν και προσπαθούμε να προτείνουμε λύσει. Οι χώρε αυτέ θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά τα κίνητρα που ήδη χρησιμοποιούν διαφορετικά. Αντί δηλαδή να δίνουν κάποιες φοροπαλλαγέ ε, εκ των προτέρων, να τις ε, παρέχουν αργότερα. Αντί δηλαδή να τις παρέχουν τοπικά, να, τι να τις συνδέσουν, να συνδέσουν τις, ε, τα, τα, κίνητρα για τους επενδυτές με μακροπρόθεσμα ωφέλη. Δηλαδή να τα συνδέσουν, για παράδειγμα, τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης αν συνεισφέρει η εταιρεία σε αυτό, θα λάβει και διάφορα ωφέλη. Έτσι ώστε να διασφαλιστεί οι εταιρείε που θα επενδύσουν πραγματικά να επενδύσουν ε, μακροπρόθεσμα, να επενδύσουν σε σχολεία, ε, σε κατάρτιση, σε, στο περιβάλλον και μετά, αφού αποδειχθεί αυτή η συνεισφορά τους, να λαμβάνουν αυτές ε, τις, αυτά τα κίνητρα. Χρειάζεται λοιπόν αλλαγή προσανατολισμού όλων αυτών των στρατηγικών ε, που δίνουν κίνητρα στους επενδυτές για τις φτωχότερες χώρες. Αυτό έχουμε προτείνει εμείς. Μας ρωτήσατε επίσης και αν οι ευρωπαϊκές συνθήκες μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο. Έχουμε κάνει μια αξιολόγηση και θεωρούμε πως εδώ έχουμε να κάνουμε με μια νέα γενιά επενδυτικών συνθήκων. Και βλέπουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη πλέον ε, τίνει να είναι η νόρμα σε αυτές τις συνθήκες και υπάρχουν ορισμένες ε, πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και λαμβάνονται ήδη υπόψη και ρυθμίζονται μέσω αυτών των ε, συνθήκων. Νομίζω λοιπόν πως δημιουργείται ένα νέο πρότυπο, ένα πρότυπο νέας γενιάς και αυτό είναι αρκετά ισχυρό. Σε πολλές περιπτώσεις ε, συνδέεται με το πλαίσιο της πολιτικής το οποίο προσπαθούμε να προωθήσουμε. Αυτό είναι το θετικό. Έγινε και μία ερώτηση για το αν το επενδυτικό δικαστήριο είναι ε, κάτι καινούριο. Εμείς θεωρούμε πως είναι ένα σημαντικό βήμα προς την μεταρρύθμιση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους. Είναι ένας ε, μηχανισμός ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα όπως είναι τώρα. Παρά το ότι έχει δώσει πολλά και έχει χρησιμεύσει. Νομίζω όμως πως χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Νομίζω πως έχετε κι εσείς την ίδια άποψη. Και χρειάζεται επίσης να δοκιμαστεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα και να διευρυνθεί αυτός ο μηχανισμός ακριβώς διότι χρειάζεται στις οικονομίες κλίμακας έτσι ώστε να παγιωθούν κάποια επιχειρηματικά μοντέλα. Χρειάζεται λοιπόν οπωσδήποτε περαιτέρω βελτίωση, όμως εμείς θεωρούμε πως είναι ένα βήμα προς τα μπροστά, προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό το είπαμε και στην Επιτροπή, το είπαμε και στα πλαίσια του ΠΟΕ, όταν παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Καναδά το κοινό τους μοντέλο αυτών των συνθήκων τον Δεκέμβριο, ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ψηφιακές οικονομίες τώρα. Για τις άμεσες ξένες επενδύσεις έχετε δίκιο. Χρειάζονται από τη μία οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. Από την άλλη όμως όλες ε, οι επενδυτικές συνθήκες ε, μέχρι τώρα έχουν αυτά τα ε, αυτές τις μικρές ερίτρες έχουν δημιουργήσει το έδαφος έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέα κοινωνικά πρότυπα, περιβαλλοντικά πρότυπα, γι' αυτό και υπάρχουν κάποια παραθυράκια. Γι' αυτό πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί. Ε, επίσης, αναφερθήκατε σε αυτή την παράλυση. Και νομίζω πως, ε, θα πατήσω λέγοντας ότι όταν λέμε προστασία των επενδύσεων, σίγουρα αυτό είναι αναγκαίο, πρέπει όμως να συνοδεύεται και από άλλες αρχές. Το δικαίωμα της ε, νομοθεσία, ε, χώρος για πολιτική, βιώσιμη ανάπτυξη, ανάληψη εταιρική ευθύνης, εταιρική διακυβέρνηση. Νομίζω πω ε, έτσι είναι μια δέσμη μέτρων αρκετά ισορροπημένη, αλλά το να δίνεις παραπάνω βάρος σε κάτι έναντι κάποιο άλλου δεν είναι σωστό. Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε και να παρακολουθούμε τις επενδύσεις που ε, και να τις προστατεύσουμε. Επενδύσεις που ε, θα έχουν στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη. Και καταλαβαίνω τις δυσκολίες που έχετε εντοπίσει στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας, αλλά εδώ νομίζω πως ε, υπάρχει προσέγγιση αυτή και προσέγγιση του συστήματος επιλύση διαφορών επενδυτή και και είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μετά διαδίκτυο για όλου. Δημόσιε ε, δημόσιες επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις. Τι πολιτική ακολουθούμε. Νομίζω πω σε μια διαφάνεια από αυτέ που είδατε αναφέρθηκε το, δημόσιο, το ενδιαφέρον του δημόσιου τομέα και το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα. Και αυτό εμείς το θεωρούμε καθοριστικό για να γίνουν αλλαγές στην οικονομία. Και νομίζω πως υπάρχει μεν έτσι, μια, κάπως, μια σύγκρουση συμφερόντων, αλλά αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αυτό είναι λίγο πολύ ε, δεδομένο. Και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να γίνει κάποια ε, αλλαγή στις, στις δυνάμεις, το ποιος είναι πιο ισχυρό Χρειάζεται επίσης να αναπτύσσουμε πάντα νέες επενδυτικές στρατηγικές και στρατηγικές ανάπτυξης. Μετά, αναπτυσσόμενες χώρες και μη. Νομίζω πως παρά την συγκέντρωση των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον ψηφιακό τομέα, που εκεί όντως παρατηρείται μια συγκεντρωτική τάση, υπάρχει τεράστιο δυναμικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες και για τις μικρές οικονομίες. Για παράδειγμα, το περιεχόμενο σε συγκεκριμένου να μέρη. Υπάρχει ένα παγκόσμιο περιεχόμενο, υπάρχει κάτι που είναι καθολικό για όλους, όμως χρειάζεται περιεχόμενο στη γλώσσα, σε μια συγκεκριμένη γλώσσα που αφορά ένα συγκεκριμένο τόπο. Και αυτό μπορεί να το δημιουργήσει μόνο μία εταιρεία που είναι βασισμένη σε αυτόν τον ε, γεωγραφικό χώρο στον οποίο θα απευθύνεται το περιεχόμενο. Οπότε αυτό στηρίζει μία ολόκληρη βιομηχανία, πολιτισμική και μη. Και νομίζω πως εδώ υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για πολλές μικρές εταιρείες σε όλο τον κόσμο και υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες ε, παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες αλλά χρειάζεται να ψηφιοποιηθούν έτσι ώστε να διαθέτουν τα προϊόντα τους και ψηφιακά. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ευκαιρίες για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις μικρές οικονομίες, τις μικρές επιχειρήσεις. Τώρα η συνεισφορά των άμεσων ξένων επενδύσεων ε, στην ποιότητα οι ποιοτικέ άμεσε ξενέ επενδύσει, ναι, συνεισφέρουν. Και με ρωτήσατε, κύριε Σόλτ, να σα αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Νομίζω το παράδειγμα τη Αιθιοπία, τη Ρουάντα και τη Ινδία είναι πολύ χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια έχουν απολαύσει τεράστια ανάπτυξη, διψήφιο, με διψήφιο νούμερο. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτό δημιουργήθηκε από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες συνεισέφεραν σε μία σε μια αύξηση 3-4%. Αυτές οι επενδύσεις ήταν κυρίως στις υποδομές, στην ηλιακή ενέργεια, στους σιδηροδρόμους, ε, σε διάφορα ε, βιομηχανικά πάρκα, κατασκευαστικό τομέα, μεταποιητικό τομέα, κλωστοϊφαντουργία, τρόφιμα και δέρματα. Είναι τομείς οι οποίοι δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, μεταφέρουν τεχνολογία, μεταφέρουν δεξιότητες. Η Ρουάντα, μέσω των επενδύσεων, ιδιαίτερα επενδύσεων στον τομέα των υπηρεσιών, προχώρησε πολύ. Λειτουργήσαμε στην ε, UNTAD συμβουλευτικά και δημιουργήσαμε και παρήχαμε μάλλον συμβουλές ε, στη Ρουάντα μεταξύ άλλων και για τον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών. Και είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Το Βιετνάμ επίσης είναι ένα άλλο καλό παράδειγμα που οι επενδύσεις οδήγησαν σε απελευθέρωση, οδήγησαν σε βελτίωση των συνθήκων. Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ναι, θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιπλέον από αυτό που κάνει, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει περισσότερες επενδύσεις που είναι φιλικές προς το περιβάλλον σε αναπτυσσόμενες χώρες, σε χώρες Αφρικής για παράδειγμα. Είναι πολύ δύσκολο να διαπραγματευτούμε τέτοιες επενδυτικές ε, συμφωνίες, οι συνθήκες, όμως αυτή την εποχή βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη αυτέ τις διάφορε κατευθυντήριε γραμμέ ε, στην πολιτική τη προσπαθεί να δημιουργήσει συνένεση ε, για νέε αρχέ που θα χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν άμεσε ξένε επενδύσει σε αυτέ τι αναπτυσσόμενε χώρε, σε αυτού του ε, τομεί που τι χρειάζονται και είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Έχετε και εσεί συνεισφέρει σημαντικά και εδώ είναι και η απόδειξη του τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Τώρα, έχουμε χρόνο ακόμα. Αν δεν έχουμε, δεν θα απαντήσω στη δική σας, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Η παρατήρηση που, έκατε, που κάνατε πράγματι είναι ε, πολύ κέρια. Υπάρχουν επενδύσεις που στόχευουν στην απελευθέρωση, ταυτόχρονα μειώνονται και οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις καθορίζονται από τρία πράγματα. Ε, πολιτική, οικονομική και κοινωνική. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη δεν είναι μεγάλη. Υπάρχει μεγάλη αστάθεια των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών, αστάθεια οικονομική, πολιτική, κίνδυνη, γεωγραφική, γεωπολιτική. Γι' αυτό και οι επενδυτές διστάζουν να επενδύσουν παρά το ότι έχουν πολλά κεφάλαια. Μάλιστα τα διάφορα ταμεία είναι γεμάτα. Δεν γίνονται επενδύσεις. Μειώθηκαν οι επενδύσεις στην Αφρική και τι κάνουμε γι' αυτό ρωτήσατε επίση. Τι γίνεται με τη διακυβέρνηση, τι γίνεται με του στόχου ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το είπα και πριν. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήσει διάφορε εταιρικέ σχέσει με αναπτυσσόμενε χώρε στην Αφρική, θα μπορέσει να μεταδώσει τι αρχέ τη, να μεταδώσει ε, αρχέ που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και να προσελκύσει καλέ επενδύσει. Τώρα, για το άλλο θέμα που με ρωτήσατε, έχουμε την μελέτη σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρατικών ε, δημοσίων διακρατικών ε, επιχειρήσεων. Το 1 τρίτο ε, του συνόλου βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κίνα έχει τις περισσότερες ως ε, μία χώρα, 200, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 400 τέτοιες επιχειρήσεις και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία και η Γαλλία που κατέχουν τις πρώτες θέσεις. εκεί οι κρατικές επενδύσεις είναι υψηλότερες, ανέρχονται στο 1,5% τον ε, του παγκόσμιου αριθμού των πολυεθνικών, όμως οι επενδύσεις ε, τους σε ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερες. Ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρ Τσάν, για αυτές τις απαντήσεις. Να μην σας χάσουμε. Το θέμα των επενδύσεων θα μας απασχολήσει το επόμενο έτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να έρθετε. Οπότε, πριν να κλείσουμε, θα ζητήσω από την Κομισιόν, εάν θέλει να σχολιάσει, ο Κάρλο Πετινάτο, επικεφαλής τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο Τζέμ Τσάν τα είπε σχεδόν όλα για τις ροές των επενδύσεων και είπε πολλά για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέκα δευτερόλεπτα μόνο για να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε υπήρξε στο προσκήνιο της μεταρρύθμισης της επενδυτικής πολιτικής από το 2010, ε, δηλαδή στην μεταρρύθμιση και των ουσιαστικών κανόνων όπως και του ε, μηχανισμού ε, διαφορών όπως αναφέρει και η έκθεση της αλλά και στη διάρκεια της δεύτερης φάσης των μεταρρύθμισης όπως την ονομάζει η UNCTAD δηλαδή της αντικατάστασης των παλαιών διμερών συνθήκων είμαστε επίσης πρωτοπόροι έχουμε ένα μέσο, ένα κανονισμό για την αντικατάσταση των διμερών συνθήκων ας πούμε η εμπορική συμφωνία με το ε, Βιετνάμ θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες συνθήκες με κάτι που θα ε, ε, περιλαμβάνει τη νέα προσέγγιση. Αυτό μας ικανοποιεί και έχει αναγνωριστεί. Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις μας εμπνέονται από το έργο της ΑΝΚΤΑΤ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Είναι πολύ ευπρόσδεκτη αυτή η δουλειά. Αυτά είχα να πω. Όσον αφορά τώρα το νέο ψηφιακό περιβάλλον, των ψηφιακών πολυεθνικών επιχειρήσεων και το γεγονός ότι όλο και λιγότερο συνδέονται με ε, φυσική παρουσία και φυσικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό είναι ένα επιπλέον επιχείρημα, όπως λέει και η έκθεση της UNCTAD. Αυτό είναι υπέρ μιας ενός ευρύτερου ε, πλαισίου πολιτικής, ε, αντί να έχουμε το κατακαιρματισμένο πλαίσιο πολιτική σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Στο σημείο λοιπόν αυτό ε, ολοκληρώσαμε τη συζήτηση του σημείου 22. Περνάμε στο 23. Και το 23 είναι η ανταλλαγή απόψεων με την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας σχετικά με τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της, ε, των προσφύγων από τη Συρία. Έχω τη μεγάλη χαρά να έχουμε εδώ τον πρέσβη μαζί μας. Καλώς ορίσατε. Και τον Ενρίκε Γκερεύο, που είναι υπεύθυνο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον εισηγητή που λείπει, αλλά η Μαρία Ελένα θα τον αντικαταστήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ε, αντικαθιστώ τον κύριο Μορέλη, ο οποίος μου έδωσε το σημείωμα το οποίο θα ήθελε να παρουσιάσει. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο συζητήσαμε εδώ το αν είναι ε, χρήσιμο να υπάρξουν κανόνες προέλευσης για κάποια προϊόντα που προέρχονται από την Ιορδανία μετά την κρίση. Παρότι ήταν συμβουλευτική συζήτηση, η περιοψηφία των συναδέλφων έδωσε την συνένεση για κάτι τέτοιο. Έτσι έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε έναν πραγματικό ενάρετο κύκλο ε, που θα ευνοήσει και τις οργανικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω του ταραχώδους περιοχής και τους 1, ε, σχεδόν 3 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία. Ένα χρόνο αργότερο ο κ. Μορέλ είναι πεπισμένος ότι αυτός ο μηχανισμός του που έχει τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο ε, είναι χρήσιμος. Υπάρχουν 15% των ε, προσφύγων που εποφελούνται από τις ε, εξαγωγές προς την Ένωση στα πλαίσια της πρωτοβουλίας όλα εκτός από όπλα. Έτσι λήφθησαν κάποιες δράσεις σε πολιτικό επίπεδο οργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 3 Μαΐου ε, σε ανώτατο επίπεδο με τη συμμετοχή της κυρίας Μάλμστρομ και του Υπουργού Βιομηχανίας της Ιορδανίας με σκοπό να γίνει γνωστό η πρωτοβουλία και έγιναν ε, στρογγυλές τράπεζες ε, από βιομηχάνους της Μεσογείου και είχε μάλλον επιτυχία. Ελήφθησαν μια σειρά από ενδιαφέροντα μέτρα όπως μια διαδικτική πλατφόρμα υποστήριξης ε, για τη δημιουργία ενός έργου αδερφοποίησης. Όσον αφορά το θεσμικό επίπεδο, χαιρόμαστε δεδομένου ότι έχουμε παρατηρητές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας, από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας στην περιοχή. Βεβαίως η πρωτοβουλία δεν λειτουργεί όσο καλά είχε προβλεφθεί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μόνο τρεις επιχειρήσεις από την Ιορδανία τις ανυποψήφιε για να χρησιμοποιήσουν τι δυνατότητε. αυτές είναι ελάχιστο. Ο κ. Μορέλ είχε την τύχη να ε, πάει πρόσφατα στο ΑΜΑΝ και οι επιχειρήσει που συνάντησε του εξέθεσαν τι τεχνικές δυσκολίε για να συμμορφωθούν με τι ευρωπαϊκέ απαιτήσει. Ζητά λοιπόν από την Επιτροπή να γίνει μια αναθεώρηση των διατάξεων, κυρίω όσον αφορά ε, περισσότερη τεχνική βοήθεια. Ενδεχομένω θα υπάρχουν κάποιε δυνατότητε βελτίωση.

είναι απαραίτητο να γίνει ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε το έργο να αποδώσει, όχι μόνο γιατί αυτό θα δώσει περιθώριο στην οικονομία τη Ιορδανία, αλλά γιατί θα βοηθήσει τι επιχειρήσει τη χώρα να απασχολήσουν περισσότερου πρόσφυγε από τη Συρία. Μόνο θετικά μπορεί να είναι ε, όλα αυτά, έτσι ώστε οι Σύριοι δεν θα θεωρούνται ανταγωνιστές των Ιορδανών, αλλά θα μπορούν να εργάζονται από τις ίδιες συνθήκες. Έτσι θα μπορέσει η Ιορδανία να δώσει περισσότερες άδειες εργασίες σε πρόσφυγες από τη Συρία, να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να δώσει περισσότερους κανόνες καταγωγής εάν αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία. Μετά με αυτό 550.000 παιδιά από τη Συρία θα μπορέσουν να πάνε σχολείο, πράγμα που αποτελεί σοβαρή πρόκληση ο χρηματοδοτικός, το χρηματοδοτικό μέσο είναι, εξακολουθεί να είναι μπλοκαρισμένο και δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις μας. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε να μας βοηθήσουν να ε, φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δώσω μέσα στο λόγο στην Κομισιόν για να μας δώσει και τη δική της οπτική. Παρακαλώ, Πετεριά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ και την κυρία Ρένα για την παρουσίαση και για τα θετικά της λόγια την πρωτοβουλία αυτή. Όπως, όπως μόλις είπε, θα γιορτάσουμε τα πρώτα γενέθλια του σχεδίου, του μηχανισμού και μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση για το που βρίσκονται τα πράγματα. Και πολύ κανά μας παρουσίασε αυτή την πρωτοβουλία. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα, αλλά όχι το μόνο τη στήριξη ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ιορδανία στο πλαίσιο τη προσφυγική κρίση και τη Συριακή κρίση. Και είμαστε αρκετά περήφανοι ω ένα καινοτόμο παράδειγμα της αξίας ε, του θεματολογίου και της δράσης τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ανταποκριθούμε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και φυσικά συνεργαζόμενοι και με την κυβέρνηση της Ιορδανίας ε, προκειμένου να δώσουμε νέα κίνητρα για τις καλές επιδόσεις της οικονομίας, να το δούμε σαν ευκαιρία παρά σαν άχθος. Η πρωτοβουλία θεσπίστηκε γρήγορα και τότε συνειδητοποιήσαμε ότι ακόμη και αν δεν εχόταν άμεσα το Κοινοβούλιο, εσείς εκφράσατε μεγάλη υποστήριξη στην πρωτοβουλία και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Όπως υπόθηκε, ισχύει αυτό το σύστημα εδώ και ένα χρόνο, θα τρέξει για 10 χρόνια και σκοπεύει να δημιουργήσει κίνητρα για οικονομική δραστηριότητα, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όχι μόνο για τους Σύρους πρόσφυγες, αλλά και για τους Ιορδανούς, που θα συνεισφέρουν στις εξαγωγές και στην παραγωγή και φυσικά θα συμβάλλει και στο να ενταχθούν οι ΣΥΡΙ στην αγορά εργασίας. Όπως υπόθηκε, έχει περάσει ένα χρόνος από την έναρξη του σχεδίου. Μέχρι τώρα ο αντίκτυπο ήταν μετριοπαθής. Δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε. Έχουμε κάπως διαφορετικά νούμερα από το ΑΜΑΝ. Μας είπαν ότι οκτώ εταιρείες έχουν εγγραφεί στο σύστημα και δύο μόνο, παρόλα αυτά δύο, άρχισαν να εξάγουν προϊόντα χρησιμοποιώντας το πλεονέκτημα αυτό της ευελιξίας που προβλέπεται στο σύστημα. 20-21 εταιρείε ε, έχουν τη δυναμική να εξάγουν υπό το σύστημα αυτό μέσα σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα και εκεί επικεντρώνουμε τις δραστηριότητές μας. Δηλαδή θέλουμε να τις υποστηρίξουμε για να το πετύχουν αυτό. Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά αριθμητικά στοιχεία, τα οποία τα εξετάζουμε τακτικά, δεν ε, υπάρχει σημαντική αλλαγή ή αύξηση στα συνολικά αριθμητικά στοιχεία. Ειλικρινά δεν το αναμέναμε αυτό πολύ γρήγορα. Και όταν ε, μιλάμε για την κατάσταση της Ιορδανίας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα ευρύτερα θέματα που πλήττουν ε, την ανταγωνιστικότητα της χώρας στην ευρωπαϊκή αγορά και την ανάγκη οι εξαγωγείς ε, να λάβουν στήριξη για να μπορούν να ανταγωνιστούν και να παρουσιαστούν εδώ στην Ευρώπη και να αναζητήσουν και να αποκτήσουν ε, μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Αναφέρθηκε το συνολικό στόχος που έχει τεθεί από την Ιρδανία να εκδοθούν 200.000 άδειε εργασία προκειμένου να ενταχθούν οι ΣΥΡΙ επίσημα στην οικονομία. Οι πιο πρόσφατε πληροφορίε που έχουμε είναι ότι περίπου 53.000 έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι οι περισσότερε από τι άδειε αυτέ σχετίζονται με τομεί όπω οι κατασκευέ ή η γεωργία όπου φυσικά δεν ε, καλύπτονται στην ε, συγκεκριμένη πρωτοβουλία των κανόνων καταγωγής όμως ε, συμβάλλουν προς την πρόοδο για την επίτευξη του συνολικού στόχου. Όπως ε, είπαμε τότε και πρέπει να αναγνωρίσουμε τώρα, η απλούστευση που προβλέπεται σε αυτό το σύστημα θέλει να δημιουργήσει πρόσθετο κίνητρο για τους οικονομικούς φορείς. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες επενδύσεις ε, στην παραγωγή ειδών για εξαγωγή στην Ευρώπη. Όμως δεν εγγυάται το σύστημα ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Δηλαδή, ότι θα έχουμε αυτές τις περαιτέρω εξαγωγέ. Αυτό εξαρτάται από την αγορά, αυτό εξαρτάται από τις δράσεις των μεμονωμένων επενδυτών, επιχειρηματιών και άλλων οικονομικών φορέων. Και φυσικά αυτοί οι οικονομικοί φορείς και επιχειρηματίες δρούν στο πλαίσιο του εθνικού κανονιστικού περιβάλλοντος στην Ιορδανία, και στο πλαίσιο της εθνικής αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη διθεσιμότητα των εργαζομένων σε συγκεκριμένους τομείς και συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Ε, όμως, ε, δεν σήκω στα χέρια ψηλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε τέλειωσε η δουλειά μας. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την Ιορδανία και το υπογραμμίζω με την Ιορδανία για να δημοσιοποιήσουμε αυτό το σύστημα, να ευαισθητοποιήσουμε διάφορους φορείς ε, και εδώ και στην Ευρώπη και να απευθυνθούμε και στην Ιορδανία σε τοπικούς φορείς και όπως υπόθηκε από την 3η Μαΐου η Επίτροπος ε, Μάλστρου μαζί με τον Υπουργό Κούντα ακριβώς οργάνωσαν ε, μία συνάντηση εδώ στις Βρυξέλλες για να δημοσιοποιήσουν ε, αυτό το σύστημα. Θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε την πρόσληψη του συστήματος, του προγράμματος, υπό αυτόν τον τρόπο και φυσικά θα κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις και στην Ιορδανία ή να χρησιμοποιούμε τα δίκτυα, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικότητας για να δημοσιεύουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Γενικά μιλώντας, ο συνολικός αντίκτυπος της πρωτοβουλίας και κατά πόσο θα αλλάξει την κατάσταση επιτόπου εξαρτάται από το επενδυτικό κλίμα στη χώρα από την ανταγωνιστικότητα των αγαθών τη Ιορδανίας στι δινέ αγορέ και στην αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο τομέα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ δεν μιλώ ως εκπρόσωπος των θεσμικών οργάνων, αλλά και για τα κράτη-μέλη και στα κράτη-μέλη αναφέρομαι, συνεργάζονται στεναρά με την Ιορδανία για να βοηθήσουν τις εταιρείε να πετύχουν αυτό το στόχο. Και επαναθετικά να αναφέρω ότι ακόμη και τρίτε χώρε όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ε, αναλάβει κάποιες τοπικές δραστηριότητες στην Ιορδανία ακριβώς για να υποστηρίξουν τις Ιορδανικές επιχειρήσεις ε, να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από αυτή την πρωτοβουλία. Τέτοια παραδείγματα, τέτοιες δράσεις συμπεριλαμβάνουν το να δημιουργούνται κέντρα απασχόλησης σε περιοχές στην Ιορδανία, προκειμένου να μπορέσουν ε, να βρουν ε, εργασιακές ευκαιρίες για Σύρους και Ιορδανούς, κυρίως στις εξαγωγικές βιομηχανίες. Και επίσης ε, αναφέρθηκε και η συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται πλήρως να υποστηρίξει την Ιορδανία στο να κάνει επιτυχία αυτή την πρωτοβουλία. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους με αυτό το στόχο και για τον ευρύτερο στόχο να υποστηρίξουμε την Ιορδανία στο να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη Συμφωνία Σύνδεσης φυσικά και για εταιρείε που δεν τυχαίνει να βρίσκονται σε αυτές τις 18 περιοχές ή να προσλαμβάνουν ένα ποσοστό σύρων προσφύγων. Τώρα, Κάτι διαδικαστικό τελευταίο. Η κοινή απόφαση του περασμένου Ιουλίου προβλέπει μια τακτική αιτήσια θεώρηση της λειτουργίας του συστήματος ε, στους ε, σχετικούς φορείς της Συμφωνίας Σύνδεσης. Μια τέτοια αναθεώρηση αναμένεται να λάβει χώρα του επόμενους μήνες βάσει μια έκθεσης που θα επιβληθεί από την Ιορδανία και θα δώσει την πρώτη ευκαιρία προκειμένου εμείς να αποτιμήσουμε από κοινού την αρχική περίοδο εφαρμογής της πρωτοβουλίας θα έχουμε διάμεση αναθεώρηση το τέταρτο έτος. Στο στάδιο αυτό πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε να λειτουργήσει η πρωτοβουλία όσο όχι αυτή τη στιγμή, παρά να ξεκινήσουμε μια διαδικασία να την επαναπροσδιορίσουμε, να την προσαρμόσουμε. Βέβαια, είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση και ευρύτερα θα θέλαμε να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε αυτή την Επιτροπή για τη διαδικασία παρακολούθηση και για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν του επόμενου μήνε. Σα ευχαριστώ για την υποστήριξή σα στην πρωτοβουλία αυτή και για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για την επιτυχία τη. Φυσικά όλοι έχουν ένα συμφέρον ε, να πετύχει αυτή η πρωτοβουλία. όμω ακούγοντά σα. στην ομιλία σα, σε 15 λεπτά, μόνο ένα νούμερο έμεινε στο μυαλό μου, ότι μόνο δύο εταιρείε χρησιμοποιούν αυτή την πρωτοβουλία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό αποτελεί επιτυχία, έτσι όλα τα άλλα μέτρα, εντάξει. Όμως ε, τελικά δεν βελτιώνει την κατάσταση. Δύο εταιρείε χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό. Είναι τρελό. Έχουμε 1,3 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Ιορδανία. Δεν είμαι ικανοποιημένο με αυτό. Ο κύριος Γκερέρο, ο ειδικό μας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή που μου δίνει το λόγο στη ζήτηση αυτή. Όχι ως γνώστη των κανόνων καταγωγής, για τα οποία ξέρω εγώ πολύ λίγο, αλλά ως μονίμου εισηγητή για την ανθρωπιστική βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και υπό το ρόλο αυτό θα πω κάποια πράγματα υπέρ της Ιορδανίας και ταυτόχρονα θα εκφράσω και κάποιες ανησυχίες για την κατάσταση των προσφύγων, κυρίως ε, των Σύρων στην Ιορδανία. Ε, μιλώντας υπέρ της Ιορδανίας, πρέπει να επισημάνουμε ότι στον κόσμο έχουμε περίπου 60 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι εκτοπισμένοι από τους τόπους καταγωγής τους. Από αυτά τα 60 εκατομμύρια, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό, περίπου 1,5 εκατομμύριο, έχει φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η ποσότητα είναι μόνο κάτι παραπάνω από τον αριθμό των προσφύγων που ζουν στην Ιορδανία. Θέλω να πω με αυτό ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μία ισοδύναμη προσπάθεια με αυτή της Ιορδανίας για την προστασία ή στο να προσφέρει στους ανθρώπους αυτούς ευκαιρίες ή υποδοχή, θα σήμαινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να δεκτεί 50 εκατομμύρια πρόσφυγες στο έδαφος της, στην επικρατειά της. Και όλη η κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, που καταστρέφει όχι μόνο τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και σχεδίου προς την ελληνική, αναφέρεται μόλις σε ένα πάρα πολύ μικρό μέρος σε σύγκριση με την προσπάθεια της Ιορδανίας. Επομένως, η χώρα αυτή έχει λάβει κατά τη διάρκεια της ιστορίας της διάφορα κύματα προσφύγων. Σήμερα στην Ιορδανία ζουν όχι μόνο οι Σύριοι πρόσφυγες, αλλά και διάφορα κύματα προσφύγων από την Παλαιστίνη ως συνέπεια των πολλαπλών πολέμων που έλαβαν χώρα στην περιοχή από το 1948 και μετά. Δεδομένες λοιπόν της προσπάθειας που κάνει η Ορδανία, νομίζω ότι έχει, έχει μεγάλο νόημα η υπογραφή του 2017 του Compact Agreement που κατά κάποιο τρόπο δέσμευε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ιορδανίας και να τις ε, δώσει κάποια σταθερότητα και εφεκτικότητα για να υπάρχει οικονομική και εμπορική πρόοδος. Όπως έχει και νόημα το ότι υποστηρίξαμε οικονομικά την Ιορδανία από την αρχή της κρίσης με 950 εκατομμύρια και 150 εκατομμύρια για ανθρωπιστική βοήθεια. Όπως έχει και νόημα η οργάνωση της διάσκεψης των δωρητών στις Βρυξέλλες για να προσφερθεί βοήθεια στην Ιορδανία. Έτσι λοιπόν, αφού κάναμε αυτή την ε, αναγνώριση στην Ιορδανία, θα εκφράσω κάποιες ανησυχίες. Εγώ επισκέφθηκα την Ιορδανία ως μόνιμος εισηγητής, πήγα στο Σατερί, στο 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Συρία, στον καταβλησμό των προσφύγων και φυσικά και στην Αμάν και μπόρεσα να δω τις δυσκολίες που βιώνει μεγάλο μέρος των Σύρων προσφύγων για να αποκτήσει άδεια εργασίας. Χωρίς άδειες εργασίας είναι αλήθεια ότι τους υποδέχονται στην Ιορδανία, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται σε μια κατάσταση αποκλεισμού εντός της Ιορδανίας και σε μια δύσκολη κατάσταση για να ξαναφτιάξουν εκεί τη ζωή τους. Επομένως, μόνο 52.000 από τους 200.000 που είχαμε ε, υποσχεθεί να λάβουν ε, αυτή την αυτές τις άδειε εργασίας. Όπως είπα, από τις 200.000 μόνο 52.000 έχουν λάβει τις άδειες αυτή τη στιγμή. Πιστεύω όμως ότι με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δώσουμε ε, μια μικρή όθηση στην ε, Ιορδανία έτσι ώστε να θεωρήσει τις ε, διαδικασίες καταγραφής και να διευκολύνει την απόκτηση αδειών εργασίας από τους πρόσφυγες. Επίσης πρέπει να αυξήσουμε την πρόσβαση σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες από την πλευρά των προσφύγων. Είτε έχουν είτε δεν έχουν έγγραφα. Γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο μέρος ε, των προσφύγων που δεν έχουν τα κατάλληλα χαρτιά. Πρέπει και να εκφράσω το εξή, επειδή είναι κοινή η θέση στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Μας ανησυχεί η διαδικασία της επιστροφής των προσφύγων στη Συρία. Ιδίως γιατί η κατάσταση στη Συρία είναι προφανώς Ίσως ε, με το πέρασμα του χρόνου σε μικρέ περιοχές της Συρίας να υπάρχουν κάποιες μικρέ περιοχές Συρίας που να είναι σίγουρες, όμως σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και επομένω κάθε επιστροφή ξαναθέτει σε κίνδυνο τη ζωή των προσφύγων που βρίσκονταν πριν στην Ιορδανία. Και υπάρχει συγκεκριμένη ενσυχία για μια ζώνη μεταξύ Συρίας και Ιορδανίας που λέγεται Ρουκμπάν. Εκεί υπάρχουν περίπου 50.000 άτομα που ουσιαστικά είναι εγκαταλελειμμένα και ακόμη και η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια είναι πραγματικά δύσκολη για τους ανθρώπους αυτούς. Συνθετικά νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την Ιορδανία. Πιστεύω ότι κάνει μια προσπάθεια που δεν μπορέσαμε να κάνουμε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να εκφράσουμε και την ανησυχία μας, ε, γιατί αφού υποδέχτηκαν τους σύρους, να μπορέσουν να τους ε, προσφέρουν συνθήκες ε, που να είναι ισότιμε με του Ιρδανού πολίτε. Αν ακολουθήσουν αυτή την οδό, νομίζω ότι η υποχρέωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να του δώσει την απαραίτητη βοήθεια για να το πετύχουν. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι λοιπόν ε, σαφές ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες είναι οι απαιτήσει. Θα δώσω όμως τώρα το λόγο και σε εσά για να μας πείτε τη δική σας άποψη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μίλησαν πιο πριν και να πω καταρχάς ότι ότι για την περιοχή αυτή υπάρχουν όντως ακόμα πρόσφυγες και η Ορδανία μαζί με τις ε, διεθνείς αποστολές των ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθεί να διευκολύνει ε, την ε, διανομή φαγητού νερού εκεί στα αναχώματα στο ΠΕΝ. Γιατί είναι τόσοι άνθρωποι εκεί. Το θέμα είναι, ασφάλι, είναι η ασφάλεια η Ορδανία, όπως ξέρετε, άνοιξε τα σύνορά της από την αρχή και υπάρχουν μέρες και νύχτες που χιλιάδες Σύριοι φτάνουν στην Ιορδανία. Τώρα τα νούμερα είναι φυσικά πολύ μικρότερα, αλλά έχουμε ανησυχίες για την ασφάλεια, διότι οι περισσότεροι από τους Σύρους σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή έρχονται από μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή, από την άλλη άκρη της Συρίας, η οποία ήταν υπό τον έλεγχο τρομοκρατικών οργανώσεων, κυρίως από το ΝΤΑΕΣ. Οι πληροφορίες λοιπόν που είχαμε σχετικά με την ασφάλεια ήταν ότι κάποιοι από εκείνους πήγαν εκεί έτσι ώστε να εκτελέσουν διάφορα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ιορδανία. Και η Ιορδανία δέχεται μεγάλες πιέσεις από τη διεθνή κοινότητα σε αυτό το στάδιο. Γι' αυτό λοιπόν ε, όταν τους ε, υποδεχτήκαμε μετά είδαμε ένα βομβαρδισμό ενός φορτηγού που είχε μέσα έξι Ορδανούς στρατιώτες και διάφορους, ε, διάφορους ε, νοσηλευτές που είχαν πάει εκεί για να βοηθήσουν τους ε, Σύρους πρόσφυγες. Μετά, θέλετε να παραμείνουν ανοιχτά τα σύνορά μας, αλλά αν το θέλετε αυτό, σας παρακαλώ να βοηθήσετε την Ιορδανία, να βοηθήσετε να αντέξουμε. Υπάρχουν χώρες γύρω μας που καταραίουν, η διεθνής κοινότητα οι εταίροι μα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μα βοηθήσουν έτσι ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τι υπηρεσίε αυτέ αυτές Σύρου. Από την πρώτη μέρα η κυβέρνησή μα, μετά από εντολή του βασιλιά έχει ανοίξει τι πόρτε τη του Σύρους και, και οι Σύροι στην Ιορδανία μπορούν να απολαύσουν όλες τι υπηρεσίες ε, που μπορούν και οι Ιορδανοί. Μπορούν να πάνε στις ε, κλινικές, τα νοσοκομεία, τα σχολεία μας, όπως ε, και οι Ορδανοί, όσο μας το επιτρέπει η χωρητικότητά μα. Τώρα υπάρχουν εκατοντάδε χιλιάδε παιδιά από τη Συρία στα σχολεία μας. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει ε, υπερφορτωθεί. Τα σχολεία δουλεύουν με δύο και, με, τρει βάρδιε τρεις βάρδιες σε πολλές περιοχές Ιορδανίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν όσο το δυνατόν περισσότερου σύρου. Η Ορδανία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και τους νέους. Όταν άρχισε η κρίση στη Συρία το 2011 και έφτασαν όλα αυτά τα παιδιά στην ε, Ιορδανία ήταν 10 χρονών. Τώρα είναι 17-18 χρονών. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια χαμένη γενιά. Αυτό είναι κακό και για την Ιορδανία και για το μέλλον της Συρίας και για την Ευρώπη. Και δεν θέλουμε αυτά τα παιδιά να πέσουν θύματα στρατολόγησης, να μείνουν εκτός σχολείου, διότι είναι πολύ εύκολο στόχος για να στρατολογηθούν από τι τρομοκρατικέ οργανώσει. Ε, για τους ε, κανόνες που αναφέρατε, ε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας. Να πω ότι ήμουν πέρυσι σε μια συνάντηση όπου συζητήθηκε αυτό το θέμα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τότε ανέφερα τις ανησυχίες της χώρας μου και ανέφερα ότι υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, υπάρχει υπάρχουν προτάσεις για συγκριτική αξιολόγηση που προτετάθηκαν από την Κομισιόν, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν και να γίνουν. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο Πρόεδρος, δεν νομίζω να καταφέρουμε τίποτα εάν υπάρχουν πολλοί προώθημοι, αλλά μόνο δύο τα κατάφεραν, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Αυτή είναι η θέλησή σας να βοηθήσετε την Ιορδανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά να, ζητούμε να χαλαρώσει κάποιες από τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας έτσι ώστε η Ορδανία να μπορέσει να εφαρμόσει τη συμφωνία και να αποκομίσει και εκείνη τα ωφέλη που θα προκύψουν από τη συμφωνία αυτή. Αυτή η συμφωνία προτάθηκε από την Ορδανία στην διάσκεψη του Λονδίνου, διότι είμαστε μια αξιόπιστη χώρα και δεν θέλαμε οι πρόσφυγες στη χώρα μας ε, να ρισκάρουν τη ζωή τους προσπαθώντας να πάνε στην Ευρώπη. Είναι πολύ πιο οικονομικό για την Ευρώπη το να μείνουν οι πρόσφυγες στην Ιορδανία. Αλλά δεν είναι μόνο χρηματικό το θέμα. Η Ιορδανία είναι και μία ενδιάμεση ζώνη ανάμεσα στη ριζοσπαστικοποίηση ε, και την τρομοκρατία προσπαθούμε και τον πολιτισμό προσπαθούμε κάθε μέρα ανταλλάσσουμε πληροφορίες ε, για τους ξένους μαχητές για τη ριζοσπαστικοποίηση προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε το σκεπτικό ήταν να οδηγηθούμε σε μία λύση με, θετικό, θετική έκβαση για όλους, αλλά τώρα ένα χρόνο αργότερα δεν βλέπουμε κάποιο όφελος για την Ιορδανία. Φυσικά ξέρουμε ότι υπάρχει καλή θέληση από τους συναδέλφους, αλλά είδαμε από την αρχή ότι αυτά τα benchmarks που έχουν τεθεί δεν μπορούμε να τα τηρήσουμε. Τώρα έχει έρθει η ώρα να σας δώσω μερικά νούμερα. Ο αριθμός των ε, επιχειρήσεων έχει αυξηθεί. Είναι 8 όπως είπατε. Δύο από αυτές ε, έχουν λάβει έγκριση και έκαναν εξαγωγές ύψους 300.000 ευρώ. Η δεύτερη εταιρεία 25.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό, των, ε, το, συνολικό, συνολικός αριθμός των ε, αδειών εργασίας τον Ιούνιο του 2017 ήταν περίπου 54.000 άδειε εργασία. Και η Ιορδανία του κυνηγά του Σύρου. κυριολεκτικά, με την καλή έννοια, και προσπαθεί να του πείσει ότι προσπαθεί, προσπαθούμε να δημοσιεύσουμε, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε, τηλεόραση, ραδιόφωνο, για να πείσουμε του σύρου, να έρθουν, να καταγραφούν, να πάρουν δωρεάν άδειε εργασίας. Αυτές οι 54.000 άδειε εργασίας εκδόθηκαν από ε, δημόσιε υπηρεσίε υπηρεσίες Ιορδανίας δωρεάν. Επίσης δίνουμε έμφαση στον πολιτισμό. Ε, εδώ έχουμε επενδύσει 32% ε, στη μεταπητικό τομέα, στην χονδρική, στην ελληνική, τις υπηρεσίες στέγασης, σύντησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί πολλοί Σύριοι πρόσφυγες έρχονται από αγροτικό από αγροτικέ περιοχές έχουν αγροτικό υπόβαθρο και θέλουν να δουλέψουν σε αυτόν τον τομέα. Προσπαθούμε λοιπόν να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, κάνουμε εργαστήρια, συνέδρια, διανέμουμε φυλάδια. Υπάρχουν πολλοί Ιορδανοί που προσπαθούν να έρθουν σε επαφές με επαγγελματικά μελητήρια, με επιχειρήσεις σε άλλες χώρες. Έχουμε διάφορα συνέδρια business to business όπως είπε και ο συνάδελφος, προσπαθούμε να διοργανώσουμε και συνέδρια σε βιομηχανικές πόλεις στην Ευρώπη, να συμμετέχουμε, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Υπάρχει όμως μια διστακτικότητα από τους Σύρους πρόσφυγες για να νομιμοποιήσουν το καθεστώς τους ως εργαζόμενοι, γιατί λαμβάνουν διάφορα μηνιαία επιδόματα, τα οποία είναι από κονδύλια ευρωπαϊκά οι Σύριοι λοιπόν που παίρνουν αυτά τα μηνύα επιδόματα δεν βλέπουν το, ρόλο για, το, το λόγο να τα χάσουν ψάχνοντας για δουλειά. Αυτό λοιπόν θέλω να τονίσω εδώ σε εσά, στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν ότι πρέπει να πάρουμε κάποια στατιστικά στοιχεία και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε αυτού του σύρου, να του μιλήσουμε και να του πείσουμε να ζητήσουν άδειε εργασία. Επίση, πολλοί Σύροι φοβούνται ότι αν καταγραφούν, καταχωρηθούν, θα χάσουν το καθεστώ του πρόσφυγα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι πρόσφυγες στην Ιορδανία από τη Συρία εργάζονται στην ε, γεωργία και σε κάποιον σχετικό τομέα και όχι στη βιομηχανία. Και παρά το γεγονός αυτό διστάζουν ακόμα και να ε, κάνουν κάποια επαγγελματική κατάρτιση. Υπάρχει επίσης ένας κατώτατος μισθός. Έχουμε 200.000 Σύρους που εργάζονται στη μαύρη αγορά πήραν αυτές τις δουλειές από ε, επιχειρήσεις ε, της Ιορδανίας και υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορούμε να δώσουμε δουλειά σε Σύρους ε, νόμιμα. Και δεν μπορούν λοιπόν να λάβουν την άδεια να εξάγουν προϊόντα. Επίση, οι βιομηχανικέ εγκαταστάσει πρέπει και εκείνε να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα για να εξάγουν τα προϊόντα του. Ε, εδώ θέλουμε τη δική σα βοήθεια. Χρειάζεται ε, βοήθεια για να δημιουργηθούν συνδέσει με του Ευρωπαίου αγοραστέ, οι οποίοι θα ε, θελήσουν να αγοράσουν τα προϊόντα της Ιορδανίας. Και το όλο σκεπτικό πίσω από αυτό ήταν να προσελκύσουμε ευρωπαϊκές επενδύσει να έρθουν στην Ιορδανία να κάνουν δουλειέ είναι αυτή τη στιγμή σχεδόν αδύνατο να γίνουν επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιορδανία, όπως γίνεται και με την Τινησία. Και παρά την καλή θέληση και των δύο πλευρών υπάρχουν πολλές προκλήσεις οι οποίες ε, καθιστούν αδύνατη, αδύνατες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Η Ιορδανία θέλει να γίνει αναθεώρηση της συμφωνίας αυτής και όταν ε, ήρθα εδώ την προηγούμενη φορά, πολλοί συνάδελφοι ε, άκουσα πω είπαν ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να είναι 20 ετή και όχι 10 ετή. Εμείς έχουμε προβλήματα. Δεν μπορούμε καν να πείσουμε τους επενδυτέ να έρθουν στην Ιορδανία για 10 χρόνια. Η αναθεώρηση λοιπόν, σύμφωνα με την ε, παρούσα συμφωνία, είναι για 5 χρόνια. Αλλά νομίζω πω ήδη ένα χρόνο μετά έχουμε δει αποδείξει ότι δεν λειτουργεί σωστά έχουμε κάποιες ενδείξεις γιατί δεν πάει καλά. Ε, μία από αυτές, και ε, μία από αυτές αιτίες είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην Ιορδανία να καταφέρουν να φτάσουν το όριο των 200.000 εργαζόμενων σύρων προσφύγων. Αυτό δεν γίνεται όπως σας έχω πει. Προσπαθούμε να τους πείσουμε συνέχεια, αλλά δεν το καταφέρνουμε και προσπαθούμε να ε, πείσουμε τις ε, επιχειρήσεις στην Ιορδανία να λάβουν την αναγκαία ε, έγκριση. Αλλά οι επιχειρήσεις δεν θέλουν να, να διαλύσουν τα εργοστάσια τους και να τα ξαναχτίσουν αλλού. Δεν έχουν αυτήν την πολυτέλεια. Νομίζω πως θα σταματήσω εδώ και θα απαντήσω σε επόμενες ερωτήσεις καθώς αυτές θα γίνουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Η κυρία Ρίση έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την κυρία Λαλόγκ. Είμαστε διάφοροι εκπρόσωποι εδώ, γιατί δεν μπόρεσε να έρθει. Θα διαβάσω τις παρατηρήσεις σας στα γαλλικά. Η κυρία Λαλόγκ, ε, χαίρεται που γίνεται σήμερα αυτή η σημαντική συζήτηση για την πρωτοβουλία αυτή, η σημαντική για την Ιορδανία και την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Είναι σημαντική, αλλά θέλει να χαιρετήσει την αλληλεγγύη και το θάρρος της χώρας, δεχόμενη στο ε, έδαφος της πάνω από 550.000 Σύρους πρόσφυγες στους οποίους προστίθενται και μια σειρά από ε, ε, πρόσφυγες από άλλες χώρες. Έχουμε το 10% σχεδόν του συνολικού πληθυσμού της χώρας και το μισό του πληθυσμού αυτού είναι παιδιά και γυναίκες. Η Ορδανία αντιμετωπίζει την ίδια πρόκληση όπως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την καταπολέμηση τρομοκρατίας και το πρόβλημα της των μεταναστευτικών ροών και δέχτηκε το, στη διάσκεψη του Λονδίνου να δεχτεί εργατικό δυναμικό. Εδώ ε, έχουμε έξι χρόνια πόλεμο που μπορεί να δημιουργήσει μια χαμένη γενιά. Η πρωτοβουλία αυτή που ζητά την χαλάρωση των κανόνων καταγωγής ε, είναι θετική για τις ε, Επιχειρήσει τη Ιορδανία. Θα ξεφύγω λίγο από τι παρατηρήσεις τη κυρία Λαλόγκ να πω αυτό που είναι ε, πολύ σημαντικό στην σημερινή απογευματινή συζήτηση. Τα νούμερα, όπως και κύριε, δώσατε κύριε εσεί, κύριε Πρόεδρε, ε, είναι ε, εντυπωσιακά. Οκτώ μόνο εταιρείε που έχουν εγγραφεί και δύο που εξάγουν και άκουσα ακόμα τις τα εντυπωσιακότερα νούμερα που έδωσε ο κύριος Πρέσβης, 25.000 ευρώ, ευρώ μιλάμε μια τεράστια ε, γενεδορία από πλευρά τη Ιορδανία και του γειτονικού Λιβάνου και ήθελα να ρωτήσω, ακούγοντα τον εκπρόσωπο τη Κομισιόν, γιατί, για ποιο λόγο υπάρχει θέμα ενημέρωση, ε, υπάρχει θέμα ανακοίνωση, διαδικασία, αλλά απήντησε ο ίδιο ο κύριο Πρέσβη. Υπάρχουν συγκριτικοί δείκτε και ε, κανόνε πρόσβαση που είναι αδύνατοι. σήμερα, μετά από ένα χρόνο, διαπιστώνουμε την σημερινή κατάσταση ε, στη συζήτηση δεν είναι ότι δεν λειτουργεί καλά, δεν λειτουργεί καθόλου το σύστημα. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε και όλοι ότι εκ μέρους της Επιτροπής μας ότι πρέπει τώρα να γίνει κάτι και θα πώς θα λύσει η Κομισιόν το πρόβλημα. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να προσφέρουμε ε, μέσα που θα είναι πρακτικής φύσεως. Επαστρέφω σε αυτά που λέει η κυρία Λαλόμ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει με στρατηγικό τρόπο την εμπορική πολιτική της για να επιδιώξει αυτούς τους αναπτυξιακούς και ανθρωπιστικούς στόχους. Έχει αναλυφθεί πρωτοβουλία, πρέπει να δοθούν περισσότερες, ε, ε, οι δυνατότητες αυτές σε περισσότερες ζώνες και πρέπει να φροντίσουμε να μην μην γίνονται απάτες και να ε, υπάρχει προτίμηση σε στοχευμένο ε, πληθυσμό και θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της ε, πρωτοβουλίας. Τις είδαμε και θα τις δούμε και πάλι. Εν κατακλείδη, θέλει να επενθυμίσει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία μας με αυτή τη χώρα σε οικονομικό και πολιτικό και αμυντικό, στον αμυντικό τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είμαι εγώ Άγγλος και έχω συνηθίσει πολύ στο αγγλικό στυλ του κυρίου ο οποίος ε, υπήρχε, υπήρχε μακροσκελής, είπε πολλά, αλλά έδωσε ελάχιστα στοιχεία. Ε, αλλά ο κύριος Λάγκε με πάρα πολύ σωστά έθεσε των δάκτυλο, επί των τύπων των ήλων. Δεν ξέρω πώς τι πρέπει να κάνουμε ότι να αποφύγουμε χιλιάδες Ευρωπαίοι γραφειοκράτες να ασχολούνται με κάτι. Και ακούσαμε νούμερα. 300.000 εξαγωγές και 25.000 ευρώ εξαγωγές. Δηλαδή τίποτα ξέρω ότι είστε κι εσείς Άγγλος, εκπλήσωμαι ότι είχατε το θάρρος να έρχετε εδώ και να μας μιλάτε επί ένα τέταρτο, επί της ουσίας για τίποτα. Ας είμαστε σοβαροί και ας δούμε το περιεχόμενο. Κοίταξα και εγώ τα νούμερα. Η Ορδανία έχει πληθυσμό περίπου 7,5 εκατομμυρίων. Το είναι λιγότερο από το 1 δέκατο του πληθυσμού της Τουρκίας. Η έκταση της Ιορδανίας είναι λιγότερο από 1 τρίτο του, της Τουρκίας. Και αν είναι σωστά τα νούμερα και μοιάζει ότι δεν ξέρω, είναι περίεργα. Το ΑΕΠ της Ιορδανίας είναι 37 δις της Τουρκίας είναι 2-3, δηλαδή 2.000 δισεκατομμύρια. Και ας δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, και πώς ε, την αντιμετωπίζεται η Ιορδανία. Η Τουρκία έχει πάρει επανειλημμένος, επανειλημμένος, επανειλημμένος χρηματοδότηση ε, πολύ μεγαλύτερη από την Ιορδανία, ενώ η Ορδανία τα αξίζει πολύ περισσότερο το σχόλιο του πρέσβη και το οποίο ε, ε, συμφωνώ Ο, ο, πρέσβης επεσήμανε ότι η ε, Ιορδανία είναι μια ρυθμιστική ζώνη και είναι λιγότερο δαπανηρό και πιο αποτελεσματικό να μην φροντίζουμε την Ιορδανία αλλά να έρθουν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λοιπόν δεν έχω καμία επιρροή αλλά αυτή τη στιγμή για ένα λεπτό σας απασχολώ και ζητώ από τα μέλη της Επιτροπής, τους Κομισιών που είναι εδώ να προχωρήσουν, να ξεφύγουν αυτό το αδιέξοδο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Σας παρακαλώ, θα πρέπει τουλάχιστον να αντιμετωπίζετε την Ιορδανία, τουλάχιστον εξίσου καλά με την Τουρκία, όσον αφορά την άμεση χρηματοδότηση. Και βεβαίως θα έπρεπε να τη μεταχειριζόμαστε ακόμα καλύτερα. Ε, υπάρχει μεγάλη διαφορά σε πολλά από τα πολιτικά ζητήματα, αλλά σήμερα ε, μοιάζει ότι ευθυγραμμιζόμαστε, ενώ συνήθως ε, έχουμε διαφορετική άποψη. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη. Δεν μπορούσα να είναι εδώ σκέδες μας σήμερα και νομίζω ότι τα περισσότερα θέματα τέθηκαν από τους συνάδελφου στην αίθουσα και οι ερωτήσεις τέθηκαν ήδη στην Κομισιόν για τα αριθμητικά στοιχεία, τις διαφορές. Ε, έτσι λοιπόν σας ευχαριστώ, αλλά Θέλω να καταγραφεί ότι το ECR αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν από την Ιορδανία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της Ιρακής κρίσης και αναγνωρίζουμε και τον αντίκτυπο στην οικονομία της Ιορδανίας και στα παραδοσιακά μοντέλα εμπορίου. Και καθώς είμαστε υπέρ να μείνουν οι πρόσφυγες ε, στην ε, περιοχή καταγωγής τους. Αγκαλιάζουμε αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι θα βελτιωθούν ε, οι συνθήκες και για τους πρόσφυγες αλλά και για, τους, ε, για τη χώρα φιλοξενίας, για τους κατοίκους. Όμως βλέπουμε ότι δεν φέρει αποτελέσματα η πρωτοβουλία αυτή και πρέπει να δούμε τι να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους πρόσφυγες που βρίσκονται επί τόπου, αλλά και να βελτιώσουμε την εμπορική ροή και τις εξαγωγές από την Ιορδανία που υποστηρίζουν τους ανθρώπους αυτούς και τις κοινότητες. Θα πρέπει όχι μόνο να έχουμε ένα έγγραφο που να λέει ότι ισχύει εκεί η πρωτοβουλία, αλλά να εφαρμόζεται, να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος θα ήθελε το λόγο. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Επομένως, Κομισιόν, ακούσατε νομίζω το σαφέ μήνυμα από όλε τι πολιτικές ομάδες και από του βουλευτές στην αίθουσα είναι πράγματι ντροπή αν συγκρίνεται το κόστος των ε, διαπραγματεύσεων το κόστος ε, του να είναι κανείς εδώ και το πόσο κοστίζουν ε, οι μισθοί των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σύγκριση με τα ωφέλη, τότε θα πρέπει να πάμε και ένα απομαντίο. Ποια είναι η στρατηγική σας για να βελτιώσετε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για το έντονο ενδιαφέρον που έδειξαν για το σύστημα αυτό. Θα Λέγα ότι ίσως ε, εγώ κάπως να μην έδωσα υπερβολική ε, έμφαση, όμως ε, ουσιαστικά πλαστικοί σωλήνες είναι αυτοί που εξάγονται στην Κύπρο και στην Ισπανία υπό το σύστημα αυτό. Αυτή είναι η μόνη εμπορική συναλλαγή που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. 300.000 ευρώ ή κάτι τέτοιο. Είναι ένας αριθμός που δόθηκε από τον πρεσβευτή, δεν θα τον... Ε, δεν θα φέρω εγώ αντίρρηση, όμως ε, πρέπει να θυμηθείτε. Ε, για περίπου 300 εκατομμύρια είναι οι εξαγωγές της Ιορδανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν έχει να κάνει με την λήψη της πρωτοβουλίας. Και Δυστυχώς ε, τώρα έχουμε τέτοια επίπεδα όπως ε, και 10 χρόνια πριν και παρόλο που δεν υπάρχουν δασμοί ε, για την πρόσβαση της Ιορδανίας στην Ευρωπαϊκή Αγορά με δύο εξαιρέσεις που είναι τα λουλούδια και το ελαιόλαδο. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε και στο θέμα της ικανότητας των Ιορδανών εμπόρων να εκμεταλλευτούν. Την κατάσταση αυτή μη χάνετε, λοιπόν την ευρύτερη εικόνα για την Ιορδανία, στο πώς μπορεί να ανταγωνιστεί στην ευρωπαϊκή αγορά, όταν εξετάζουμε την συγκεκριμένη πρωτοβουλία που πήραμε εμείς για τους κανόνε καταγωγής πριν 12 μήνες. Όπως σας είπα, περιμένουμε την ευκαιρία να κάνουμε την πρώτη αναθεώρηση του συστήματος. Άκουσα κάποια στοιχεία τώρα από τον πρεσβευτή που δεν τα είχα ξανακούσει. Έτσι λοιπόν περιμένουμε την πρωτογραπτή έκθεση από την Ιορδανία που θα δώσει μια νέα ζωή σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι εμποδίζει τις εταιρείε ε, να εκμεταλλευτούν το σύστημα ή τους επενδυτές να έρθουν στην Ιορδανία και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα. Και όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ανοιχτό μυαλό τρόπο. Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της πρωτοβουλίας, ε, ήταν αποτέλεσμα έξι μηνών εργασία μεταξύ Ιορδανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήταν δηλαδή ιδιαίτερα μακροστελής διαπραγματεύσεις. Ακολούθησε μια πρόταση που έγινε το Δεκέμβριο του 2015 από την Ιορδανία και αυτή περιοριζόταν στο να επιτρέψει να εργαστούν οι ΣΥΡΙ πρόσφυγες σε 4-5 συγκεκριμένες περιοχές ε, της χώρα και κατόπιν της ενθάρρυνσης της Κομισιόν διευρύναμε αυτές τις ε, περιοχές και καταλήξαμε στο να απελευθερώσουμε τους κανόνες καταγωγής για όλα τα βιομηχανικά προϊόντα Βέβαια, ο δεσμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη μηδενικό, δεν έχει σημασία που είναι ο προτιμησιακό κανόνα καταγωγή. Όμω, εκεί που υπήρχε ένα κεφάλαιο ότι ελάχιστοι, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, είχαν δυνατότητα σε προτιμησιακούς κανόνες ε, καταγωγής. Αυτό ίσχυε και για την Ιερδονία και εμείς Κομισιόν προτείναμε να το θέσουμε επιτάπητος και το βάλαμε στην απόφαση. Αυτό που δεν κάναμε ήταν τότε να μιλήσουμε για απελευθέρωση από τους κανόνες καταγωγής για τα αγροτικά προϊόντα. Αν ένα προϊόν ε, δεν καλλιεργείται εκεί επιτόπου ή δεν αλλιεύεται επιτόπου στην Ιορδανία, σημαίνει ότι πρέπει να εισαχθεί πριν τη μεταποίηση. Αυτό είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο επομένω, ένας πολύ πιο πολύπλοκος τομέας και θα είμαι μαζί σας. Δεν θέλαμε και αυτή είναι η όλη λογική της πρωτοβουλίας, βασίστηκε στην ιδέα στο να μπουν οι Σύριοι πρόσφυγες στην επίσημη αγορά εργασίας. Ήδη δουλεύουν, άτυπα πιστεύουμε. Θέλαμε λοιπόν ε, να τους ε, φέρουμε στην επίσημη αγορά εργασία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν σύμβαση, άδεια εργασία, θα πρέπει να περάσουν μια κυβερνητική διαδικασία. Για κάποιους από τους πρόσφυγες αυτό ίσως να είναι πρόβλημα, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερη ευελιξία για κάποιου άλλου ε, οικονομικούς ε, παραγόντες ε, μπορεί να είναι πρόβλημα γιατί σημαίνει μεγαλύτερη τυποποίηση. Εμείς απ' έξω δεν μπορούμε να καθορίσουμε τις συνθήκες της αγοράς εργασίας. Πρέπει να εργαστούμε με όλα όσα υπάρχουν διοικοί. και όπως σας είπα, περιμένω την ευκαιρία να δούμε, από την Ιορδανία, στην επόμενη αναθεώρηση για το αν υπάρχουν συμφορήσεις στο σύστημα, αν μπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές αλλά όπως είπα στην εισαγωγή μου, πιστεύω ότι οι αλλαγές θα χρειαστούν επίσημη νομοθεσία από την πλευρά μας. Έτσι όπως χρειάστηκε για να υλοποιήσουμε το σύστημα. Και αυτό χρειάζεται φυσικά χρόνο. Υπάρχει λοιπόν και ένα ευκαιριακό κόστος εδώ να ξεκινήσουμε από το μηδέν ή να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε θεμελιώδη στοιχεία του συστήματος. Αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε. Αυτά θα έλεγα εγώ για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα σχολιάσω α, όσους μίλησαν για τη γενικότερη σχέση με την Ιορδανία, όμως χτες ήμουν σε ένα συμβούλιο σύνδεσης και η Ιορδανία ήταν πολύ θετική σε σχέση με το επίπεδο υποστήριξης που δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ιορδανία. Φυσικά, σε ένα πολύ πιο συγκεκριμένο πλαίσιο όπω αυτό, είναι εύκολο να δούμε που είναι τα ελλείμματα. Αλλά νομίζω πρέπει να έχουμε κατά νου και την ευρύτερη εικόνα. Πάντως, σας ευχαριστώ πολύ το ενδιαφέρον της Επιτροπής σας για την πρωτοβουλία αυτή. I've got a point of order. Έχω κάτι διαδικαστικό να πω. Την τελευταία εβδομάδα είχα πολύ χρόνο, φαίνεται, και μου φαίνεται κάπως παράξενο και ακατάλληλο, αν θέλετε, και κάτι που εκδηλώνει ασέβεια από μέρους της Επιτροπής, ότι δεν κάνει την παραμικρή προσπάθεια να απαντήσει στις πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Μάλιστα τις ε, προσπέρασε έτσι βιαστικά και θα ήθελα να καταγραφεί αυτό. Ναι, ε, να, για να είμαι ειλικρινής δεν ήταν διαδικαστικό θέμα αυτό. Αλλά, κύριε Πρέσβη, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Πράγματι, σε πολιτικό επίπεδο, στο υψηλότερο επίπεδο, υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις. Υπάρχει ένα ε, συμβούλιο σύνδεσης πολύ επιτυχημένο τώρα πρόσφατα χθε. Υπάρχει όμως και συμφωνία σύνδεσης και, ανάμεσα στην Ιορδανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της είναι να στηριχθεί οικονομική ανάπτυξη στην Ιορδανία και το εμπορικό ισοζύγιο ανάμεσα στην Ιορδανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ορδανία εξάγει περίπου 200-300 εκατομμύρια ε, ε, ευρώ σε προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει προ την Ιορδανία πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν ποιο αποφελείται σε αυτή την περίπτωση. Και βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση τώρα, σε μια θέση που μας έχει φέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις διαπραγματεύσεις για τη Νέα Συμφωνία. Ε, αυτό βέβαια είναι ένα επιπλέον πρόβλημα που δημιουργείται και με τους ε, τόσο πολλούς Σύρους πρόσφυγες. Οι, μη, οι Ορδανοί είναι ε, αρκετοί. Είναι περισσότεροι από ό,τι συνηθίζεται. Έχουμε πάνω από 50.000 ε, Λίβιους και Ιεμενίτες πέρα από τους Σύριους. Μετά, Υπάρχουν ορισμένοι χριστιανοί και ε, γεσίντοι από μέρη του Ιράκ που διώκονται θρησκευτικά και το μόνο ασφαλές μέρος για εκείνους είναι η Ορδανία. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πήγαν στην Ορδανία, απολαμβάνουν ξεθρησκεία ανεξάρτητα από το θρησκευτικό τους ε, παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για να συνοψίσουμε λοιπόν θα δώσω το λόγο στη Μαρία Ρενά. Ε, νομίζω ότι ομόφωνα σχεδόν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει, μπας περιπτώσει, να μην περιμένουμε να αναθεωρηθεί η διάταξη που, ε, όπως προβλέπετε για το 2020, ε, υπάρχει μια συγκεκριμένη διατύπωση και ο κύριος Μορέλ ζήτησε ε, η αναθεώρηση να γίνει όσο το πιο γρήγορα για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αντίθετα άκουσα κάποιες ομιλίες εδώ στο πλαίσιο της Επιτροπής μας. Κάποιοι επιτίθεται στην Κομισιόν για έλλειψη αποτελεσματικότητα ε, του μέσου αυτού και είναι οι πρώτοι που λένε ότι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν τους μετανάστες στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει μία οικονομία που μπορεί να ενσωματώσει τους πρόσφυγες, είναι η ευρωπαϊκή οικονομία. Θεωρώ λοιπόν ότι εκ μέρου κάποιων είναι λίγο υπερβολικό να επιτίθεται στην Κομισιόν για τη μία αποτελεσματικότητα ε, του μέσου, ενώ όταν μιλάμε για την κατανομή και την υποδοχή των ε, προσφύγων στην Ευρώπη είναι οι πρώτοι που αρνούνται. Άρα μπορούμε πολύ καλά να πούμε ότι υπάρχει έλλειψη σήμερα αποτελεσματικότητας η οποία δεν οφείλεται κατά ανάγκη στο, ε, ε, στην μη αποτελεσματικότητα της Κομισιόν αλλά τη δυσκολία να δουλέψουμε πάνω σε τέτοιες μηχανισμούς, σε τέτοιες σημαντικές διατάξεις αλλά α σταματήσουμε να είμαστε υποκριτέ, οι οποία καμιά φορά κυριαρχεί σε αυτό το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται ε, το σημείο 23 και θα παρακολουθήσουμε το θέμα. Θα είμαστε σε στενή επαφή με την Κομισιόν για να δούμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες ώστε να έχουμε καλύτερες αναφορές του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Τώρα, θέμα 24 είναι, θεωρώ πιο ευχάριστο, δεδομένου ότι αφορά τα αλκοολούχα ποτά, The labeling. την, ε, τις ενδείξεις, την επισήμανση και τις γεωγραφικές ενδείξεις, την προστασία μάλλον των γεωγραφικών ενδείξεων. Είναι ένα ευχάριστο θέμα. Έχουμε εδώ τον εισηγητή, τον Νίκολα Ντάντι, στον οποίο και θα δώσω τον λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος ε, στόχος της πρότασης κανονισμού που συζητάμε σήμερα είναι η ευθυγράμμιση της ε, ισχύουσα σχετικής νομοθεσίας με τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και το Εξουδότης τη και εκτελεστικέ Αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως ε, πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τροποποιεί ορισμένα ουσιαστικά στοιχεία του κανονισμού του 2008 και εισάγει νέα στοιχεία με πιθανή επίπτωση σε τομείς αρμοδιότητας της δικής μας Επιτροπής. Ο στόχος των ε, τροποποιήσεων είναι λοιπόν, των τροπολογιών είναι διατηρήσουμε τουλάχιστον το επίπεδο προστασίας που έχει η σημερινή νομοθεσία όπως ε, ήδη έχει υποθεί στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων συζητάμε για ένα τομέα των αρκολούχων ποτών που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς των ευρωπαϊκών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων και περιλαμβάνει προϊόντα υψηλής ε, αξίας ε, γιατί είναι παραδοσιακά προϊόντα και πρώτες σύλλες που αναφέρονται σε πολύ συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, οι γεωγραφικές ενδείξεις αποτελούν το κατάλληλο εργαλείο για την προστασία του διακριτικού χαρακτήρα και της ποιότητας των προϊόντων. Αυτά έχουν γίνει ένα από τα μεγαλύτερα επιθετικά συμφέροντα της κοινή εμπορική πολιτικής μέσω του οποίου προσπαθούμε να πετύχουμε ένα ανάλογο επίπεδο προστασίας με το ευρωπαϊκό και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ε, τρίτων, ε, στις αγορές των τρίτων χωρών. Έτσι λοιπόν θα ήταν καλό να αναπτύξουμε ένα όσο περισσότερο ομοιόμορφο πλαίσιο των γεωγραφικών ομπασιών, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα διάφορων τομέων. Αυτό θα ενισχύει την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο στο θέμα αυτό και ιδίως στις διαπραγματεύσεις των εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες όπως όλες οι μορφές δικαιωμάτων ε, διανοητικής διοκτησίας και οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να είναι θύμα καταχρήσεων και γι' αυτό ε, θα ε, πρέπει να ενισχύσουμε την προστασία από την παραχάραξη και τις δόλες πρακτικές. Ε, στις τροπολογίες έχουμε την πρόταση να αναπτυχθεί μια νομοθεσία που να επιτρέψει την εμπλοκή και την, ε, το σταμάτημα των παραποιημένων γεωγραφικών ε, ενδείξεων τα οποία περνούν από έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φτάσουν σε τρεις χώρες. Οι υπόλοιπε τροπολογίες αναφέρονται σε συγκεκριμένα στοιχεία του κανονισμού που έχουν να κάνουν με τις δικές μας αρμοδιότητες. Συγκεκριμένο, καταρχήν, το πρώτο θέμα αφορά ε, την μετάφραση των ονομάτων στην ετικέτα. Πρέπει να έχουμε μια διάταξη που να προβλέπει την ιδιότητα για τα αλκαλούχα ποτά που προορίζονται για εξαγωγή, να αναγράφεται στην ετικέτα πέρα από την πρότυπη ονομασία της γεωγραφικής ένδειξης και η μετάφρασή της και σε άλλη γλώσσα, πέρα από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αυτό απαιτείται, από την νομοθεσία ενός τρίτου κράτους. Αυτό το στοιχείο είναι ουσιαστικό για τις εξαγωγές. Το δεύτερο σημείο αφορά το ηλεκτρονικό μετρό και τα χαρακτηριστικά του. Το ηλεκτρονικό μητρό θα πρέπει να είναι ένα διαφανές δυναμικό εργαλείο προσβάσιμο που να έχει την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα 3 του κανονισμού 110-2008 θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτόματα τις γεωγραφικές ενδείξεις που καταχωρίζονται και προβλέπονται στο παράρτημα και η Κομισιόν θα πρέπει να τις επαληθεύει όταν μπαίνει σε ισχύ ο νέος κανονισμός. Θεωρώ πολύ σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται και οι γεωγραφικές ενδείξεις ε, των τρίτων χωρών και να προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Διεθνή Συμφωνία. Αν το επιθυμούν οι τρίτες χώρες ε, βέβαια. Έτσι λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των εμπειρικών διαπραγματεύσεων με τις τρίτες χώρες. Κάποιες χώρες από την Μερκοσούρη ήδη έχουν δηλώσει ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Το τρίτο σημείο αφορά ε, ουσιαστικά το χρονοδιάγραμμα. Η καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται σε ένα κατάλληλο χρονικό πλαίσιο. Προτείνω να πάμε από τους 12 στους 6 μήνες ε, το χρόνο εξέτασης. Αυτό έχει να κάνει με τα καθεστώτα των διατροφικών προϊόντων. Έτσι θα έχουμε ουσιαστικά και ομοιόμορφους χρόνους. Και το τελευταίο σημείο έχει να κάνει με την ε, χορήγηση και το συζήτηση της ερμοδιότητες. Ε, εδώ προβλέπεται καθορισμένη περίοδος 5 ετών με δυνατότητα παράτωσης για περίοδος αυτής της διάρκειας. Όμως, καθώς εδώ μιλάμε για ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού, θεωρείται απαραίτητο το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να αξιολογήσουν ε, τα αποτελέσματα ε, έχοντας ε, κατά νου τον αντίκτυπο στους επιμέρους τομείς. Αυτές είναι οι σκέψεις για τις τροπολογίες που έχω παρουσιάσει και εγώ θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια καλή δουλειά στο θέμα αυτό και να παρουσιάσουμε μια γνωμοδότηση χρήσιμη και για τη δουλειά των άλλων συναδέλφων στις Επιτροπές Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Προτείνετε και οι δοκιμές. Θέλω να δώσω καταρχήν το λόγο στους γεώδεις συζητητές. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, όπως πολύ σωστά είπατε, μετά την ε, παρατεταμένη συζήτηση του προηγούμενου θέματος, καλό είναι να ε, αισθανθούμε λίγο καλύτερα με την μεθυστική προοπτική αυτή τη έκθεση. Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να, την, ε, να πω ότι είναι απολύτω ευπρόσδεκτη η πρόταση για τη βελτίωση των ε, υφιστάμενων κανόνων στον τεχνικό αυτό τομέα, τον ορισμό τη προστασία και τη σήμανση των αλκοολούχων ποτών, συμπεριλαμβανομένων και των γεωγραφικών ενδείξεων. Και παρότι ο προτινόμενο ε, κανονισμός ε, αλλά είναι πολύ διαφορετικό πιστεύω ότι είναι κατάλληλος για το τομέα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχει ε, ε, ε, επανέλθει η αρχική αγροτική η νομική βάση. 95% αυτών των ποτών πηγαίνουν σε 80 διεθνείς αγορές. Αν φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο θα αφαιρέσει το σκοτσέζικο ουίσκι από τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ενδιαφέρον. Ενώ το κείμενο της ευθυγράμμης αφορά τον κανονισμό και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη ε, διαδικασία καταχώρησης των προϊόντων αυτών, των αλκοολούχων ποσών, αυτό αλλάζει και πολλά άλλα πράγματα. Χαίρομαι που δεν σκοπεύει η Κομισιόν να εισάγει αλλαγές στις πρακτικές παραγωγής. Τις περισσότερες ε, περιπτώσεις οι αλλαγές που προτείνει η Κομισιόν δεν προκαλούν ανησυχία. Όμως κάποιες ε, προσαρμογές, ε, οι διορθώσεις ληστική φύσεως θα μας επιτρέψουν να μην έχουμε προβλήματα. Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις η πρόταση εισάγει νέες αλλαγές πολιτικής που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά εμπορικά προβλήματα και πρέπει να τα μας απασχολήσουν. Θέλω να ε, πω ότι είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση του συναδέλφου Νικόλα Ντάντη για κάποιες αλλαγές. Έχω μελετήσει διάφορες τροπολογίες, οι περισσότερες από τι οποίε θέλουν να αφαιρέσουν τις συγκρούσεις από τις δυσκολίες με την νέα διατύπωση, να διορθώσουν λάθη ή να ε, ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα. Επίσης κάποιες προσπαθούν να επιλύσουν τις σοβαρότερες δυσκολίες που εισάγει η να ξεκαθαρισουν ορισμενα πραγματα επισης καποιες προσπαθουν να επιλυσουν τις σοβαροτερες δυσκολίε που εισαγει η προταση και αφορούν τη διευκρίνηση του Μητρώου του νέου ε, τελωνιακού κώδικα και όλα τα θέματα της παραχάραξης ε, των δόλιων πρακτικών που ε, στοιχίζουν στην, κοινο, στην Ένωση 4,3 δις. Η σημασία όλου αυτού είναι σημαντική όταν θέλουμε να επιμείνουμε ε, στις μελλοντικέ εμπορικές διαπραγματεύσεις, κυρίως με τις, ε, στην Νοτιοανατολική Ασία, όπου υπάρχει τεράστια δυνατότητα για εξαγωγές. Ευχαριστώ. Thank you, I can agree with... Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με πολλά από τα σχόλια που έκανε ο κ. Κέλλη. Το Brexit και το whisky, εντάξει είναι θέματα, αλλά πέραν αυτών αναγνωρίζουμε και εμείς την ευρύτερη δομή ως πιο κατάλληλη αλλά μας ανησυχεί η επάρκεια κάποιων διατάξεων που θα διασφαλίσουν το επίπεδα προστασίας και τις ε, εμπορικές ελευθερίες. Χαιρόμαστε τουλάχιστον, όπως είπε ο εισηγητής, ε, με τις ε, νέες εισαγωγές και τις τροπολογίες σχετικέ με αυτό. Καθώς και με τις τροπολογίες που αφορούν την ανάγκη να ακούσουμε τις ανάγκες του τομέα. Χρειάζεται λοιπόν ε, να ληφθούν υπόψη όλες οι επιτυχίες των ε, εξαγωγών που είναι πάνω από, 2, ε, από 10 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν το 50% αυτού του όγκου του εξαγωγών. Πρέπει να διασφαλίσουμε η νέα πρόταση να μην δημιουργήσει νέο διοικητικό άχθος και να μην θέσει σε κίνδυνο τις εξαγωγές και καλωσορίζουμε τις τροπολογίες που θα επιφέρουν ασφάλεια δικαίου στο ηλεκτρονικό μήτρο που θα αντικαταστήσει το παράρτημα 3 της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και την επανεισαγωγή της ε, δυνατότητας ε, της ε, μετάφρασης χωρίς να χρειαστούν πράξεις καταξιδότηση από την Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τα παραποιημένα προϊόντα άσχετα από τον προορισμό τους και τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να κλείσει το κενό στην υφιστάμενη νομοθεσία και να χρησιμοποιήσει μια πολιτική που θα είναι πιο αποτελεσματική, θα προστατεύει τα εμπορικά σήματα και ε, θα φροντίζει έτσι ώστε να ε, αναγνωρίζονται τα πλαστά εμπορικά σήματα και να ε, απομακρύνονται από την αγορά. Θεωρούμε πως μπορεί να υπάρξει επαρκής προστασία υπό εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν ποιο θα χρησιμοποιήσουν. Δεν θεωρούμε όμως πως υπάρχει ανάγκη για αυτήν τη συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 22. Σε γενικέ γραμμές όμως θεωρούμε ότι ο, ο έκανε πολύ καλή δουλειά και θα χαρούμε στην συνεργασία μαζί του και με τους υπόλοιπους κοιόδες για να βρούμε μια συμβαστική λύση και ένα καλό μπαρ για να τα απολαύσουμε όλα αυτά τα ποτά. Ευχαριστώ πολύ. Η Φεντερίκα, εκ μέρους των Φιλελεύθερων. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε εξαντλητική αντιληπτική απόψεων. Ήδη η πρώτη εξαντλητική απόψεως ήταν χωρίς έγγραφο. Νομίζω ότι είναι γνωστές όμως οι θέσεις ε, των διαφόρων. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τη δουλειά του. Και από τη δική μου πλευρά τα ουσιαστικά πράγματα εδώ είναι να εξυγχρονίσουμε τη διαδικασία καταχώρησης των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται στην Ευρώπη με τρεις πρωταρχικούς στόχους. Να ενισχύσουμε την προστασία, να αυξήσουμε την νομική ασφάλεια είναι ουσιαστικό για τους παραγωγούς μας και μας το λένε συνεχώς και να ενημερώσουμε καλύτερα τους καταναλωτές. Το σχέδιο έκθεσης φυσικά οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση και ευχαριστώ τον εισηγητή ο οποίος ε, εδώ αναφέρει μια σειρά θεμάτων που συζητήσαμε το Μάιο. Νομίζω ότι το ουσιαστικό που εκφράστηκε είναι το εξή. το νέο ηλεκτρονικό μητρό για να έχουμε ασφάλεια δικαίου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί πρέπει να πλουστευτεί η διαδικασία καταχώρησης και να είναι προσβάσιμες στον καταναλωτή όλες οι πληροφορίες με διαφανή τρόπο. Επίσης, η δυνατότητα μετάφρασης των γεωγραφικών ενδείξεων στη γλώσσα της ε, τρίτης χώρας όταν το απαιτεί η νομοθεσία εκεί για να μην ποινικοποιήσουμε τις εξαγωγικές αγορές μας. Επίσης, ε, οι αγορές που παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση, πάνω από 5% για την Κεντρική και Νοτιοαμερική, Αμερική, περίπου 5% για την Αφρική και τη Μεσανατολή και πάνω από 4% για την Ουσία, είναι σημαντικό. Και είναι και μια ανησυχία που συζήτησαμε πολλού συναδέλφου. Δηλαδή, θέλουμε να ζητήσουμε προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων να εφαρμοστεί και στα αλκοολούχα που είναι σε διέλευση από την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Είναι ουσιαστικό για να καταπολεμήσουμε την παραποίηση που κοστίζει 140 εκατομμύρια το χρόνο και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι όλα αυτά θα βρεθούν στο τελικό κείμενο μετά την ψηφοφορία. Ωστόσο, το είπα και το Μάιο και θα το επαναλάβω. Δεν ε, θα εκπλαγώ για το ότι βλέπω εδώ μία σιωπή για την επέκταση των εκτελεστικών πράξεων που προτείνει η Κομισιόν. Θέλω να είμαι σύντομη και να μην πω σε τεχνικά ζητήματα, Πρόεδρε, και θα πω το εξή. Νομίζω ότι το σημερινό κείμενο δίνει λευκή επιταγή στην Κομισιόν, η οποία στο μέλλον θα μπορεί να δεκτεί ή να αρνηθεί ή να καταργεί την καταγραφή των γεωγραφικών ενδείξεων, χωρίς να μπορούμε εμείς να φέρουμε κάποια αντίρρηξη. Άκουσα τα επιχειρήματα του εισηγητή, ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ε, ικανότητα αντίδρασής μας. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αιτιολογεί να εγκαταλείψουμε την δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου του που έχουμε. Έτσι λοιπόν θα βάλω μια τέτοια τροπολογία για να περιορίσω τις εκτελεστικές πράξεις όπως ε, σας είπα και τελευταία φορά, ε, εγώ είμαι μέλος και στην Επιτροπή Προπολογισμού και η κυρία Γιούσο εκεί, που είναι η συγγήτρια, θα καταθέσει μια παρόμοια τροπολογία για τις εκτελεστικές πράξεις. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο προϊόν ε, εξαγωγής, πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε αξία, επομένως είναι κάτι πολύ φιλόδοξο για μας και νομίζω ότι τελικά μπορούμε να βρούμε και μία συνεννόηση. Ευχαριστώ πολύ. Για τους πράσινους, κύριε Φορέντζα. Όχι, για τους πράσινους, για την Κούα, συγγνώμη. Ναι, δεν άλλαξα ομάδα. Και εμείς ε, ως GUNGL ε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την γνωμοδότηση. Και εμείς είμαστε υπέρ της ε, πρωτοβουλίας που παίρνει η Κομισιόν. Προφανώς η προτεραιότητά μας παραμένει να βελτιώσουμε το επίπεδο προστασία για έναν τόσο σημαντικό τομέα όπως αυτή των αλκοολούχων ποτών ένα τομέα που πρέπει να υποστηριχθεί στο να διατηρήσει υψηλό επίπεδο παραγωγή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο προς αυτή την κατεύθυνση που θα συνεισφέρει στο να διατηρήσουμε αυτή την παραγωγή στην επικράτεια και να εγγυάται τα δικαιώματα των καταναλωτών και μια διαφανή και Στην ουσία του κειμένου έχουμε κάποια σημαντικά στοιχεία εμείς ε, δεν ε, συμφωνούμε ε, με την δευτερογενή νομοθεσία που προτείνει η Κομισιόν, γι' αυτό θέλουμε να χρησιμοποιηθούν εκτελεστικές πράξεις και κατεξουσιοδότηση πράξης, περιορίζοντας τον περιορισμό παρέκκλησης από τον κανονισμό όταν μιλάμε για ουσιώδη στοιχεία της πρότασης. Επίσης, θέλουμε η δυνατότητες, οι αρμοδιότητες να ισχύουν για μία περίοδο όχι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια. Ε, θα πρέπει ουσιαστικά να γίνεται η μετάφραση της ετικέτας ε, χωρίς να δίνεται έγκριση της Κομισιόν. Θεωρούμε ότι είναι γραφειοκρατικό και δεν βλέπουμε αυτή την αναγκαιότητα. Συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι η καταπολέμηση της παραχάρηξης είναι κάτι πολύ σημαντικό στο πεδίο αυτό η ευθύνη ελέγχου ότι οι πρωτοστατευόμενε γεωγραφικέ ενδείξει δεν χρησιμοποιούνται παράνομα ε, ανήκει στα κράτη-μέλη και η Κομισιόν πρέπει να ενημερώνεται για την εφαρμογή των κανόνων. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα κατάλληλο πλαίσιο που να επιτρέπει να αποσυρθούν από την αγορά τα παραποιημένα ποτά. Ε, Επίση πρέπει να αποφευχθούν ε, κάποιε παρεξηγήσει για τον καταναλωτή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το εμπόριο με τρίτες χώρες. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ξεκαθαρίζουμε τους κανόνες διαδικασίας του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μητρώου για αυτό το τύπο, προ... Ε, για αυτό το τύπο ποτών αποτελεί πρόοδο, είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους μικρούς παραγωγούς ε, και μπορεί να ε, τους επιτρέψει να επιβιώσουν και να έχουν αξιοπρεπή ζωή. Αυτό το μητρό θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό. Οι κανόνες ουσιαστικά πρέπει να είναι κατανοητοί και στους παραγωγούς. Ευχαριστώ. Η Τιτσιάνα Μπεγκίν για το EFTD. Ευχαριστώ. Εμεί στην ε, Ιταλία και στην Ευρώπη παράγουμε πάρα πολύ υψηλής ποιότητας ε, αλκαλούχα ε, ποτά 150 εκατομμύρια παραξία παράγουμε στη χώρα μας. Έχουμε 38 αλκοολούχα ποτά που παράζουμε στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν ευχαριστώ τον συγητή για το κείμενο αυτό το οποίο πρέπει ουσιαστικά να τροποποιήσει το νομικό πλαίσιο δυνάμει τη συνθήκη της Λισαμβόνας. Εγώ συμφωνώ με το ότι ε, θα έχουμε μετάφραση της ετικέτας σε τρίτες ε, χώρες και το γεγονό ότι θα ισχύει ουσιαστικά θα έχει την ίδια νομική αξία το Μητρό με τον κανονισμό 110. Ο εισηγητής ε, βέβαια ε, παρουσίασε τα στοιχεία από τη σκοπιά του διεθνούς εμπορίου. Όμως ε, θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν γιατί υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για τη γενική πρόταση και φυσικά αυτό έχει και αντίκτυπο και στην εμπορική πτυχή. Καταρχήν, Κάποιε αμφιβολίε για το άρθρο 8, παράγραφος 5 δηλαδή, για την ε, διάταξη σε σχέση με τι αρωματικέ ουσίε ε, που μιμούνται προστατευόμενα από τα Παραδείγματο χάρη, εδώ πιστεύω ότι αυτή η παράγραφος ε, μπορεί να θέσει σε εμπορία εκτός της Ένωσης ποτά που αντιγράφουν ε, το πρωτότυπο και είμαστε στα όρια της ε, παραχάραξης και της νοθείας. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν στο άρθρο 38 διάλεξε τις κατεξουσιοδότηση πράξη για τον περιορισμό των γεωγραφικών ζωνών. Αυτό θα πρέπει να γίνεται διαφορετικά. Είναι συμβατό λοιπόν λοιπόν αυτό το άρθρο με την αρχή της επικουρικότητας και σε σχέση με το άρθρο 34 δεν βλέπω μια ποια αιτιολόγηση Κομισιόν ε, μπορεί να ακυρώσει μια γεωγραφική άνοιξη μέσω εκτελεστικών ε, πράξεων. Εδώ ε, αυτό θα πρέπει να είναι επιλογή του κράτους προέλευσης, όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο εισηγητής έχει τροποποιήσει αυτό το άρθρο 19 για μια συγκεκριμένη περίοδο. Επίση, κατανοώ ότι χρειάζεται επικαιροποίηση, όμω νομίζω ότι η Κομισιόν πηγαίνει μακριά και αναλαμβάνει αρμοδιότητες που θα έπρεπε ουσιαστικά να επιμεριστούν με τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να μας δώσει λεπτομερέστερη εξήγηση για το γεγονός ότι πρέπει, πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ομοιομορφία στην Ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Μάρτιν από τη Ευχαριστώ πολύ. να έχουμε κι εμείς ε, έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Όσον Κέλλη ε, έκανε πολύ ένα, καλό ένα πολύ καλό σχόλιο για το Brexit. Δεν νομίζω πως το εμπόριο και οι εμπορικές διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μείωση των δασμών, θα προστατεύσουν το σκοτσέζικο, το ιρλανδικό ουίσκι. Δυστυχώ ε, δεν είναι καλά να είναι το σκοτσέζικο ουίσκι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκολα για την πολύ καλή δουλειά όμω που έκανε. Δύο είναι οι ανησυχίε μου. Σχεδόν δύο. Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει να ακολουθήσουμε τους κανόνες της Τελωνιακής Ένωσης εάν θέλουμε να έχουμε μία τικέτα επισήμανση προέλευσης. Δεν νομίζω πως αυτοί οι κανόνες του τελωνιακού κώδικα είναι κατάλληλοι σε αυτήν την περίπτωση. Γιατί, γιατί, ας δούμε το σκοτσέζικο ουίσκι, που είναι πραγματική περίπτωση και πουλά στη Γαλλία ουίσκι, ας πούμε, από τέσσερα διαφορετικά αποστακτήρια. Τα φέρνει σε αυτά τα ποτά στη Γαλλία, τα αναμειγνύεις. Σύμφωνα με τους κανόνες ε, προέλευσης, αυτό θα είναι προϊόν Γαλλίας. Από την άλλη, αν πάρει σκοτσέζικο ουίσκι, το στείλει στη Βουλγαρία, του προσθέσει διάφορε αρωματικέ ουσίε, το προϊόν αυτό, παρότι θα αποτελείται από 85% σκοτσέζικο ουίσκι, θα θεωρείται προϊόν Βουλγαρίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε, δεν θα είναι λογικό τον τελωνιακό κώδικα. Και μια άλλη ανησυχία, λιγότερο σημαντική, στις αιτιολογικές σκέψεις, ο Νίκολα έχει εισαγάγει μια διάταξη για να αποφτράψει την διέλευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων, ε, προστατευμένων προϊόντων. Νομίζω πως έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε γενικές γραμμές και τον ευχαριστώ για την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης ε, Γεωργίας και Εμπορίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε από τη Γενική Διεύθυνση Αγκρή και ε, ο συνάδελφος που είναι επίσης ε, από την Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Ε, μιλάμε όμως με την ίδια φωνή με την Γενική Διεύθυνση Trade. Θα του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ο παραγωγικός διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρόσθετος μετά την έγκριση της πρότασης της Κομισιόν της την 1η Δεκεμβρίου 2016 ο τομέας των αλκοολούχων ποτών προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στο γεωργικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι στρατηγικής σημασίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ο κανονισμός του 2008 για τα αλκοολούχα ποσά λειτουργήσε καλά στο παρελθόν και παρήχε σημαντική ανάπτυξη στον τομέα. Η πρόταση της Κομισιόν δεν επιδιώκει την αλλαγή των κανόνων αλλά βελτίωση του νομοθετικού κειμένου και απλούστευση την, τις ε, τρέχουσες διαδικασίες γεωγραφικών ενδείξεων που είναι μακροσκελείς και δυσκίνητες. Γι' αυτό ε, ε, χαιρετίζει τις τροπολογίες του αξιότιμου Ευρωβουλευτή του κυρίου Τάντι και ο οποίος έχει τους ίδιους στόχους και φέρει πολύτιμες βελτιώσεις στο κείμενο. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες από πλευράς Κομισιόν για κάποιες από αυτές τις τροπολογίες, κυρίως στο κομμάτι που αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις. Παραδείγματο χάρη, το θέμα του μήκους, της διάρκειας τη, του ελέγχου της Κομισιόν, η προθεσμία των έξι μηνών για τον έλεγχο το, της εφαρμογής της γεωγραφικής ένδειξης είναι ευαίσθητο θέμα και πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά. Πριν υποστηρίξουμε μια τέτοια δέσμευση πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι αρμόδιες επιτροπές, ε, υπηρεσίες κομισιών είναι σε θέση να τηρήσουν αυτή την προθεσμία. Αν παραδείγματο χάρη ο κανονισμό, σύμφωνα με την αρχή τη επικουρικότητα, θα μπορούσε να καθορίζει τον έλεγχο της αίτηση ως ανεπαρχή κυρίως λόγω της ευθύνης του κράτους μέλους, όπως ισχύει στην περίπτωση του τομέα των τροφίμων, παραδείγματος χάρη, αυτό θα επηρεάσει θετικά τη διάρκεια του ελέγχου της Κομισιόν. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να καλύπτει την ευρωπαϊκή διάσταση, παραδείγματος χάρη, να κάνει τις ε, ε, αντιρρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά η αξιολόγηση θα γίνεται κυρίως σε επίπεδο κράτους μέλους και η Κομισιόν θα κάνει έναν απλό έλεγχο ότι δεν υπάρχουν προφανή λάθη. Μια τέτοια προσέγγιση θα επιτρέψει τον έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πραγματοποιηθεί σε συντομότερο διάστημα. Επιπλέον, υπάρχει τροπολογία για τις αιτιολογικές σκέψεις που απαγορεύουν την, ε, τους κανόνες της γεωγραφικής ενδείξης για ε, προ, προϊόντα που βρίσκονται σε, ε, που διέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό μοιάζει ότι είναι ασυνεπές. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κανόνας που να σχετίζεται με αυτή την αιτιολογική σκέψη. Το θέμα της συστηματικής αντικατάστασης με τον όρο προστατευμένη ε, πριν από τη γεωγραφική ένδειξη με τον όρο καταχωρισμένη είναι κάτι που θα πρέπει να ε, ε, συζητηθεί. Νομίζω ότι η Κομισιόν επιδιώκει το πιο ικανοποιητικό και ισόρροπο αποτέλεσμα που επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα του αλκοολούχου πορτών και γι' αυτό είναι διατεθειμένη ανα πάσα στιγμή να εξηγήσει και να συζητήσει οποιαδήποτε θέματα που μπορεί να είναι ασαφή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μιλήσατε με μια φωνή. Για να, δώσω το... να κλείσουμε το θέμα, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ντάντη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης και όλους τους άλλους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Δυνάμει των παρεμβάσεων ε, και των ε, σκέψεων που προτάθηκαν, δεν ε, θα υπάρξει δυσκολία στο να καταλήξουμε σε κοινή λύση και να έχουμε μια ωραία γνωμοδότηση που να βρίσκει όσο δυνατόν περισσότερους σύμφωνους. Ίσως να μην ήμουν πολύ φιλόδοξος ε, και ε, λυπάμαι γι' αυτό σε σχέση με την οθία και την παραχάραξη. Γιατί απλώς ε, θέτουμε ένα, μια τηλεοκή σκέψη στην αρχή, ο David G της ε, τροπολογία και εγώ θα ζητήσω να μπει στο διατακτικό αυτή τη λογική σκέψη και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε βελτίωση και σε αυτό το θέμα. Σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν, προβλέψαμε να έχουμε το ίμιση του χρόνου από 12 σε 6 μήνες, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένας ε, ομοιογενής κανόνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζονται βέβαια έξι μήνες ε, για την ανάλυση και για να γνωριστεί η γεωγραφική ένδειξη για ένα τυρί. Νομίζω ότι οι έξι μήνες μπορεί να χρειάζονται και για ένα αλκοολούχο ποτό. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει αν έχουμε ομοιόμορφους χρόνους, αν θέλουμε για ένα προϊόν έξι μήνες, γιατί για ένα άλλο να θέλουμε δώδεκα. Έτσι λοιπόν ζητούμε από την Κομισιόν να κάνει όλους τους ελέγχους πριν από τη θέση σε ίσχυ του κανονισμού και η επικαιροποίηση του πλαισίου των αλκοολούχων που θα μπουν στο Μητρό να γίνει πριν από τη θέση σύσχη του κανονισμού για να μην υπάρχουν επικαλύψεις ή δυσκολίες. Πιστεύω ότι αυτά τα στοιχεία βρίσκουν σύμφωνος και τους συλλαδέλφους. Σας ευχαριστώ όλους και περιμένω τις τροπολογίες σας. Πιστεύω ότι με αυτέ θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε περαιτέρω το κείμενο. Ο Πρόεδρο ε, μας κάλεσε και για ευσυγνωσία. Εγώ συμφωνώ και θα πρότεινα στο τέλος της συνεδρίασης κάποιος συνάδελφος να φέρει και μια φιάλη έξω από την αίθουσα και ίσως θα δούμε αν είναι καλύτερο το σκοτσέζικο ουίσκι ή το ιρλανδέζικο ουίσκι της ε, συναδέλφου του συναδέλφου Κέλλη που θα φέρει από τη χώρα του. Ο καθένας μας ε, βέβαια μπορεί να φέρει κάτι από τη χώρα του για να δοκιμάσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Perfect, Τέλειο. Τέλειο. Θα δούμε λοιπόν τι είδο η γεωγραφικής προέλευσης ε, αλκοολούχου ποτό θα έχουμε. Η έγκριση λοιπόν της έκθεσης θα είναι στις 25 Σεπτεμβρίου. Προσέξτε, 25 Σεπτεμβρίου γιατί θα, γίνει, θα δοκιμάσουμε πολλά ε, αλκοολούχα ποσά από όλη την Ευρώπη. Προθεσμοί υποβολή ε, τροπολογιών 14 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε τις διαφορετικές αρμοδιότητες των διαφόρων επιτροπών, την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΝΒΙ και ΙΝΤΡΑ, έτσι ώστε να μην έχω την ε, χαρά να ε, λέω ότι κάποιες τροπολογίες είναι απαράδεκτες. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το σημείο 24. Φτάνουμε στο 25 και 26. Είναι η σύσταση σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αυστραλία και αντιστοίχως με τη Νέα Ζηλανδία. Ο η συγγητή είναι ο Ντάνιελ Κασπάρη. Του δίνω το λόγο ευθύ αμέσω. Αγαπητά κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ήδη συγκεντρώσει μεγάλη πλειοψηφία και έχουμε ήδη συζητήσει πολλές φορές ε, για να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Γι' αυτό λοιπόν ε, στην τελευταία εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έγιναν πάρα πολλά. Έγινε μία διερευνητική άσκηση, ένα scoping exercise, το οποίο νομίζω πως ήταν προς ε, όφελος και των δύο πλευρών, προτού την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Και ε, αναμένουμε στη διάρκεια του έτους και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η, να, λά, να λάβει τη διαπραγματευτική εντολή και για την Αυστραλία και για την ε, Νέα Ζηλανδία. Η δική μας Επιτροπή έχει ζητηθεί να συντάξει μια έκθεση και μετά θα προχωρήσει το θέμα στην Ολομέλεια. Έχουμε μια πρόταση για ε, σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Έχουν αναφερθεί πολλά θέματα τα οποία μας ε, απασχολούν το σημαντικό είναι να δημιουργηθεί πρόσβαση στην αγορά της Αυστραλίας και της Νέας Ιλανδίας, να βελτιωθεί ε, ο τομέας των δημόσιων συμβάσεων, να δημιουργηθούν προοπτικές χωρίς να υποβαθμιστούν τα πρότυπα και χωρίς περιορισμούς από διάφορες ε, πτυχές εμπορικής δραστηριότητας. Ε, επίσης, δεν ξεχνάμε τους, τον τομέα του πολιτισμού. Δεδομένων τούτων, λοιπόν, κατάφερα να συντάξω ένα σχέδιο έκθεσης που Νομίζω πως ε, τα συμπεριλαμβάνει αυτά. Υπάρχουν ωστόσο αρκετές, ε, αρκετά σκοτεινά σημεία, αρκετά σαφή σημεία. Γι' αυτό λοιπόν δεν είμαι σίγουρος για τις τροπολογίες. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να τις εξετάσουμε ε, πριν περάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο διαπραγματευτικής εντολής. Αλλά υπάρχουν και συνάδελφοι από τις άλλες επιτροπές οι οποίοι θα έπρεπε και εκείνοι να συνεισφέρουν, να πούν τις απόψεις τους. Ε, μιλάμε για τις συνδεδεμένε επιτροπές, η Επιτροπή Γεωργίας θα γνωμοδοτήσει και μαζί ζήτησε αρκετό χρόνο, νομίζω πως θα έπρεπε να τους τον δώσουμε. Αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο προγραμματίζει να ολοκληρώσει το θέμα αυτό στις 10 Νοεμβρίου. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας ε, μετα ε, βάσει την ε, πρότασή της εγκαίρως, έτσι ώστε να μπορέσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί πριν αποφασίσει το Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε να μας παραδώσουν την ανακοίνωση εγκαίρως. Και γιατί ζητούμε εμπορικές σχέσεις. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι πολύ σημαντική εταίροι, όχι μόνο ιστορικά, αλλά είναι και ε, πολύ επίκαιροι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που μπορούμε να ε, βελτιώσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις, τις οικονομικές μας σχέσεις, ε, να συμπληρώσουμε τις ήδη πολύ καλές σχέσεις μας με ακόμα περισσότερα προϊόντα, με το αρνίσιο κρέας για παράδειγμα ή Νέα Ζηλανδία είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος, ε, γιατί μπορεί να μας στέλνει αρνίσιο κρέας μια διαφορετική εποχή του χρόνου, κατά την οποία δεν ε, μπορούμε να το προμηθευτούμε στην Ευρώπη. Γι' αυτό υπάρχουν λόγω γεωγραφίας ε, πολλά ωφέλη που θα έρθουν με το άνοιγμα των εμπορικών σχέσεων με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Υπάρχουν όμως πολλές δυσκολίες, υπάρχουν πρότυπα, για παράδειγμα, μία αναγνώριση προτύπων, τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν είτε μέσω δασμών είτε ε, μέσω άλλων ε, μεθόδων. Υπάρχουν λοιπόν πολλά εμπόδια αυτή τη στιγμή τα οποία θα μπορούμε να παραμερίσουμε με μια τέτοια συμφωνία και πρέπει εμείς να κάνουμε ε, ό,τι μπορούμε και να διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή θα εργαστεί με μεγάλη προσοχή αλλά και γρήγορα έτσι ώστε να προλάβουμε μέχρι το τέλος του έτου να έχουμε, να έχουμε μια απόφαση. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Η σιωπή των αμνών λοιπόν δεν θα πρέπει να μας απασχολεί τόσο πολύ να ανοίξουμε εμπορικές σχέσεις με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, Κάρολιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα σιωπήσω σαν αμνός, αλλά έχω πολλά να πω. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή και για τα δύο σχέδια έκθεσης. Συμφωνούμε ότι χρειάζεται μια δίκαιη συμφωνία με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και θέλουμε μια συμφωνία από την οποία να μπορούν να υποφεληθούν όλοι οι πολίτες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην επαναλάβουμε τα λάδι του παρελθόντος, αλλά να μάθουμε από αυτά, να μιλήσουμε για τους ε, προβληματικούς ε, τομείς και να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία η οποία θα είναι καλή και θα αποτελέσει υπόδειγμα για μελλοντικές συμφωνίες. Γι' αυτό Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί κυρώσεων στο κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα στην συμφωνία και στις δύο συμφωνίες μάλλον. Εάν έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία με αυτές τις δύο χώρες, νομίζω πως ε, θα δώσουμε το καλό παράδειγμα και για επόμενες ε, συμφωνίες. Μου λείπουν κάποια σημαντικά σημεία στην ε, έκθεση, όπως σας είπα, το κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα. Στο, ψήφι, στο σχέδιο εδώ δεν αναφέρεται και αναρωτιέμαι γιατί. Διότι πέρυσι ψηφίσαμε από κοινού ένα ψήφισμα το οποίο ζητά να υπάρξει κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα Θα υποβάλουμε και άλλες τροπολογίε, για παράδειγμα για την κοινωνική εταιρική ευθύνη, για τη, τα ε, πρότυπα του, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και για τη σύσταση διάφορων συμβουλευτικών ε, ομάδων όπως αναφέρθηκε επίσης έναν μηχανισμό κυρώσεων για το κεφάλαιο βιωσιμότητας. Μετά υπάρχουν σημεία όπως η διαφάνεια, η ρυθμιστική συνεργασία, αλλά και ε, να αναγνωρίσουμε τον ευάλωτο χαρακτήρα της ε, γεωργίας που χρειάζεται ασφαλιστικές δικλείδες, διασφάλιση το, τη των ε, υπηρεσιών αποφυγή της ε, φοροδιαφυγής, καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Αυτή είναι το στους οποίους θα υποβάλουμε τροπολογίες. Επίσης, να αναφερθώ λίγο στο, στη συμφωνία με την Σιγκαπούρη για την, ε, και, για την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Εδώ θα υπάρξει κάποιος μικτός χαρακτήρας ή θα έχουμε μια ξεχωριστή συμφωνία για τις επενδύσεις και μια ξεχωριστή συμφωνία εμπορικών συναλλαγών. Επίσης, ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χωρίσει αυτές τις ε, δύο ε, συμφωνίες, αυτά τα δύο μέρη. Εμείς καταφέραμε να οδηγηθούμε σε μια κοινή θέση. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια λύση στο δυνατόν γρηγορότερα. Ήδη έχω συνομιλήσει με αρκετούς ε, εκπροσώπους από την Αυστραλία οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για το ποιο δίκαιο θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που θα προσφύγουμε σε μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Υπάρχει μια πρόταση από εμάς πρώτα να χρησιμοποιήσουμε και να εξαντλήσουμε τα εθνικά ένδικα μέσα προτού προσφύγουμε σε επενδυτικό δικαστήριο. Μετά παρατήρησα ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 15η Σεπτεμβρίου. Νομίζω πως είναι αρκετά φιλόδοξη η σεπτεμβριου νομιζω πω ακριβώς γιατί ακριβω γιατι μετά τι θερινέ διακοπέ. Και όπω είπε και ο κύριο Κασπάρη, η διαπραγματευτική εντολή θα ψηφιστεί από το Συμβούλιο στα τέλη του έτου. Μετά θα πάμε με την αντιπροσωπεία και την Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία στι χώρε αυτέ και νομίζω πω θα ήταν καλό να έχει γνωμοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Γεωργίας πριν. Γι' αυτό και θα πρέπει να τους καλέσουμε να συμμετέχουν ενεργά. Ελπίζω να έχουμε αρκετό χρόνο για να προλάβουμε, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος χωρίς να έχει γίνει πρώτα μια αρχική ανταλλαγή απόψεων. Βλέπω πως βιαζόμαστε πάρα πολύ και πως κινδυνεύουμε να χάσουμε την αναγκαία ποιότητα που πρέπει να έχει αυτή η πρόταση. Οι διαπραγματεύσει, όπω είπε και ο Ντάνιελ Κασπάρη, πρέπει να είναι ε, χαρακτηρισμένε από διαφάνεια, πρέπει να τηρούνται τα ε, διεθνή πρότυπα και να προσπαθήσουμε να δώσουμε επίσης μια ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν, να διατηρήσουμε τα εργασιακά δικαιώματα, να υπάρχει κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα, να συμπεριληφθεί η κοινωνία των πολιτών και ε, τέλος, θα ήθελα να πω πως είμαι σίγουρη για το ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω ξανά τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Την, ε, στην πρώτη συνεδρίαση μετά τις ελληνές διακοπές θα επανέλθουμε για να δούμε τι έχει γίνει και πώς έχει κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν είναι και απόλυτη αυτή η ημερομηνία. Μην βιάζεστε, να δούμε πρώτα και τι θα κάνει το Συμβούλιο. Προσωρινά όμως η προθεσμία υποβολή τροπολογιών θα καθοριστεί στο τέλος Αυγούστου. Ο Ντέιβιντ Κάμπελ ή έμαθε το λόγο. Λοιπόν, είμαστε δύο στη τιμή του ενό ECR ε, σήμερα, γιατί έχουμε χωρίσει την ανάθεση Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Θα κάνω κάποιε γενικέ παρατηρήσει για την Αυστραλία και κατόπιν ο Ντέιβιτ ε, για την Νέα Ζηλανδία. Θέλω όμω να συγχαρώ τον εισηγητή για την πρωτοβουλία και ελπίζω ότι αυτά τα ψηφίσματα θα παρακινήσουν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις το φθινόπωρο. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι εταίροι με τους οποίους συμφωνούμε, έχουμε, κοινές, έχουμε δεσμούς και κοινούς, κοινές προσεγγίσεις, όπως επίσης και το διαμοιρασμό του ελεύθερου και ανοιχτού εμπορίου. Είναι σημαντικό να, έχουμε, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με την Αυστραλία. Έχουμε μια εμπορική σχέση, η οποία είναι ισχυρή. Το διμερές είναι 70 δις το 2016. Ε, Οι δυνατότητες της ε, σχέσης αυτής μένουν ανεκμετάλλευτες σε μεγάλο βαθμό και μια ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα το αντιμετώπιζε αυτό. Είναι καθυστερημένη. Η Αυστραλία έχει τέτοιου είδους συμφωνίες με πολλούς από τους εμπορικούς εταίρους και έχει ενσωματωθεί όλο και περισσότερο στις ασιατικές αγορές που είναι στρατηγικές. Η ομάδα μου στηρίζει το ψήφισμα για την, ε, τη σύσταση για την ε, ε, Αυστραλία και προσβλέπει την βελτιωμένη ε, πρόσβαση στην αγορά και την κατάργηση των ε, δασμολογικών και μη δασμολογικών ε, εμποδίων. Ταυτόχρονα υπάρχουμε, έχουμε μια πραγματική ευκαιρία. Καθώς κοιτάμε τον παγκόσμιο στίβο πρέπει να είμαστε τολμηροί, γρήγοροι και να, να ανταποκριθούμε με το, στο, σε αυτό που μας πρόσφεραν οι Αυστραλοί και να ολοκληρώσουμε το ταχύτερο δυνατόν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Προσβλέπουμε στην ολοκλήρωσή και εγώ είμαι το άλλο μισό της όλης ε, πράξης αυτής. Ε, ε δύο καπέλα. Είμαι σκιώδης εισηγητή ε, στο θέμα τη Νέα Ζηλανδία. Επαναλαμβάνω αυτά που είπε η συνάδελφο για τη σημασία τη Νέα Ζηλανδία ω εταίρου. Η φυστάμενη συμφωνία, η διμερή συμφωνία για την ε, αναγνώριση κάποιων τεχνικών πιστοποιητικών και η κτηνιατρική συμφωνία ε, αποτελούν μια ισχυρή πλατφόρμα επί τη οποία μπορούμε να χτίσουμε μια βαθύτερη και ισχυρότερη εμπορική σχέση και νομίζω ότι το μοντέλο θα προσωμιάζει με αυτό του Καναδά, τη ΣΥΤΑ για την Αυστραλία και την Ιαπωνία. Ε, και η Νέα Ζηλανδία έχει ένα διαφανές και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρά τα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χάνει μερίδιο αγορά στην αναπτυσσόμενη αυτή αγορά. Ε, έχουμε μειωθεί, έχει μειωθεί κατά 4% στο, η συμμετοχή μας στην συναλλαγή της χώρας και αυτό θα συνεχίσει αν δεν αλλάξει η ε, σχέση μας. Ε, Συμμεριζόμαστε τις απόψεις του ε, εισηγητή και πιστεύουμε ότι μέσω της Νέας Ζηλανδίας θα μας επιτρέψει να επεκταθούμε στις αγορές Ασίας, θα μας εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις παντός μεγέθους θα υποφεληθούν. Επιπλέον η Νέα Ζηλανδία έχει καταναλωτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για την καινοτομία και την τεχνολογία όπως οι ηλεκτρονικές μέθοδοι πληρωμής και η έξυπνη τεχνολογία. Ε, ε, πιστεύουμε ότι θα ενισχυθεί η αγορά και θα προσφέρουν ευκαιρίες σε αυτούς που ε, βρίσκονται στην αιχμή τη τεχνολογίας. Η ECR λοιπόν πιστεύει ότι θα ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή η Κομισιόν και θα διαπραγματευτεί μια φιλόδοξη συμφωνία. Ευχαριστώ. Εκ μέρου του κοιτών Φιλελευθέρων, ο κύριος Τάκουλα hatulla. Eli liberaalien ja Oliko, oliko what about uh, my heavenly language, the Finnish? Do we have anyone who is... Uh, Τι γίνεται με τα φιλανδικά, λέει ο μιλητής. So, no, yeah. Ξέρετε γιατί είναι μια γλώσσα. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω τα κακά αγγλικά μου. Καταρχήν ε, θέλω να πω ευχαριστώ στον Πρόεδρο. Εμείς ε, έχουμε μόνο ένα ρόλο, ένα καπέλο το, την Αυστραλία και την Ζηλανδία ταυτόχρονα τα συζητάμε αυτά τα θέματα. Όμως ε, προσπαθούμε να δούμε ότι το κόκκινο κρασί να έρχεται από την Αυστραλία, το άσπρο από την Νέα Ζηλανδία. Τέλος πάντων, ευχαριστώ τον κύριο Κασπάρη για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Είναι αδύνατο για μένα να βρω κάτι να διαφωνήσω για το θέμα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Είναι και οι δύο πολύ σημαντικοί εμπορικοί εταίροι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι αυτές οι συμφωνίες θα δώσουν νέες δυνατότητες σε ευρωπαϊκές εταιρείες ε, και ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας. Νομίζω ότι η συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης με του Αυστραλού επιχειρηματίε πριν δύο εβδομάδες μας ε, έδωσε μια καλή επισκόπηση του μεγάλου αριθμού των τομέων στους οποίους μπορούμε να έχουμε πολύτιμη συνεργασία. Υπηρεσίε, ηλεκτρονικό εμπόριο και επενδύσεις θα είναι σημαντικά κεφάλαια τη συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι ο Ντενίλ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα στο σχέδιο της έκθεσης και νομίζω ότι έχει θίξει όλα τα σχετικά σημεία. Μέχρι τώρα μόνο να συμφωνήσω μπορώ να ζήσω, αλλά αν βρω κάτι με το οποίο διαφωνώ θα στο γνωστοποιήσω. Και δεν υπάρχει και φιλανδική διερμηνία και έτσι με υποχρεώνει ο πρόεδρος να μακρηγορώ. Μάλιστα, να είστε ακριβείς και σύντομος. Φυσικά μπορείτε να καταθέσετε τις τροπολογίες σας στα φιλανδικά, κανένα πρόβλημα. Για την ΚΟΕ, η κυρία Μινέρ. Μπορώ να μιλήσω Ολλανδικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συγητή. Έχουμε μια... Δεν υπάρχει αντίρρηση επί της αρχής για τη συμφωνία με αυτές τις ε, δύο χώρες. Κοιτάξτε, αν πρόκειται και προϊόντα που δεν μπορούσαν ε, να παραχθούν αλλού, να το σκεφτούμε. Αλλά αν μιλάμε τώρα για προϊόντα που ταξιδεύουν όλο τον πλανήτη για να έρθουν εδώ να τα παράγουμε κι εμείς, γιατί, γιατί να εισαγαγούμε μαζικά γάλα από την Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, ενώ έχουμε κι εμείς, παραδείγματος χάρη, αγελάδες. Και ακούσαμε διάφορους όρους λόγους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τα λοιπά. Όμως ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο ένα και διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες και εδώ δεν εξυπηρετούμε την επιτευξή των στόχων της ε, Συμφωνίας του Παρισιού. Το αντίθετο. Ουσιαστικά αυτές οι συμφωνίες ε, καταπολεμούν ε, τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Η Αυστραλία όμως ε, δεν είναι καλός ε, μαθητής. Ο Καναδάς ούτε αυτός σέβεται το κλίμα τώρα για τη διατησία. Ξέρω ότι έχει ε, μία συμφωνία με την Κίνα η Αυστραλία και αυτό μπορεί να θέσει πρόβλημα. Τώρα, αν η Κομισιόν επιμένει για αυτές τις ε, ιδιωτικές ε, διατησίες, ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες που έχουν συμβάσεις ιδιωτικής διατησίας και αυτό δεν είναι τόσο καλό όσο θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Η Αυστραλία είναι κράτος δικαίου. Γιατί λοιπόν πρέπει να έχουμε τέτοιες ιδιωτικές διατησίες Επήρχε στην Αυστραλία ε, μαζικές διαδηλώσεις κατά μιας νομοθεσίας που στρέβλωνε τον κώδικα εργασίας. Έτσι λοιπόν πρέπει η Κομισιόν να είναι προσεκτική και σε αυτό, να μην υπάρχει διάλυση των κοινωνικών κανόνων. Ε, ελπίζω ότι θα μας δώσετε το κείμενο το συντομότερο για να μπορούμε να το εξετάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Για τους πρασίνους ο κύριος Μπούχνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να συμφωνήσω και εγώ με αυτά που είπε η κυρία Μινέρ και να ρωτήσω επιπλέον γιατί και αυτές οι δύο συμφωνίες ε, μοιάζουν τόσο πολύ. Οι χώρες αυτές είναι πολύ διαφορετικές η μία με την άλλη. Και νομίζω πως ε, αν έχουμε κατά νου τα προϊόντα τα ίδια πρέπει να αναγνωρίσουμε ορισμένες διαφορές. Το πιο σημαντικό σημείο για εμένα εδώ είναι η περίπτωση της Νέας Ζηλανδίας. Πέρα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που θα ε, ακολουθήσουν, αληθεύει ότι η Νέα Ζηλανδία μπορεί να ε, παράγει φθηνότερα αγαθά. Εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς, πρέπει να συνεχίσουμε ε, να ε, να σκεφτόμαστε όλες τις πτυχές, να δούμε, τι να δούμε το καλό των ζώων, να, δούμε, να συγκρίνουμε τι, πώς παράγουν στη Νέα Ζηλανδία και πώς ε, παράγουν οι κτηνοτρόφοι στην πατρίδα μου, στη Βαβαρία ας πούμε, να δούμε ποιες είναι οι τάσεις. Εδώ πρέπει δηλαδή να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτά που κάνουμε, ενδεχομένως χωρίς να ξέρουμε. Όπως είπε και η κυρία Μινέρ, για εμάς Υπάρχει ένα μεγάλο ε, πρόβλημα με τον άνθρακα. Υπάρχει ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας το οποίο τροφοδοτείται με άνθρακα από την Αυστραλία και αυτό το εργοστάσιο παράγει περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα από ότι όλη η συνολική κυκλοφορία οχημάτων στο Μόναχο. Μόνο αυτό. Εδώ λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε τι γίνεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Και οι δύο αυτές συμφωνίες νομίζω θα είναι πολύ διαφορετικές εάν υιοθετήσουμε και αυτή την διάσταση. Ευχαριστώ πολύ και η κυρία Μπεγκίν τέλος για την EFTD. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κασπάρη για το έργο του την ε, διαπραγμάτευση μια συμπορική συμφωνία με την Αυστραλία και Νέα δεν θα έπρεπε να είναι κάτι επίμαχο. Έχουμε παλιέ και παγιωμένε εμπορικέ σχέσει με τι χώρε αυτέ, όμω έχουμε κάποια ευαίσθητα σημεία για το περιβάλλον, όπω ανέφεραν ε, οι συνάδελφοι, αλλά και στον τομέα τη γεωργία. Ε, Παραδείγματο χάρη, οι τομεί τη γεωργία και του περιβάλλοντο μπορεί να πλητούν ε, αρνητικά. Έτσι λοιπόν πρέπει να μετριάσουμε τον αντίκτυπο στους παραγωγούς μας, ε, κυρίως σε όσους παράγουν κρέας, ε, τυριά και δημητριακά. Πέρα από αυτές τις δυσκολίες θα πρέπει να είναι εκτός ο δρόμος. Όπως είπε ο εισηγητής, πρόκειται για δύο χώρες που σέβονται πλήρως το κράτος δικαίου υπάρχει ασφάλεια δικαίου και προστασία των επενδυτών. Και ακριβώς γι' αυτό δεν συμφωνώ με την επιμονή της Κομισιόν που θέλει με κάθε κόστος ε, να εντάξει εδώ το περίφημο ε, σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων. Ξέρουμε ότι δεν τη θέλουν οι εταίροι μας, έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει εδώ να δούμε ότι στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία ε, οι πολίτες ε, δεν θέλουν ε, αυτή τη ρήτρα, ούτε οι Ευρωπαίοι πολίτες τη θέλουν. Το Συμβούλιο θα έπρεπε τουλάχιστον να θέσει στην δική μας διάθεση το κείμενο για να δούμε ποια θα είναι η διαπραγματευτική θέση της Ένωσης. Και τέλος, δεν πιστεύω ότι είναι καλό να διαιρέσουμε στα δύο κάποια συμφωνία για να αποφύγουμε την ψηφοφορία των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αντίθετα, πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και να τους επιτρέψουμε να εκφραστούν επί το σύνολο της συμφωνίας. Αυτή είναι η δική μας θέση. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν θα πω ότι η διαπραγματευτική εντολή πρέπει να είναι διαθέσιμη μόνο στου ευρωβουλευτέ. Όχι, η διαπραγματευτική εντολή πρέπει να είναι ε, δημόσια προσβάσιμη, έτσι ώστε ο καθένα να μπορεί να διαβάσει περί τίνο πρόκειται. Ο Πέτερ Μπέρτ είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα σχολιάσει αυτά που συζητήσαμε. Αλλά το κεντρικό μου ερώτημα είναι πότε θα έχουμε ένα σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χαίρεται που ήρθε γέρος και το έχει επικοδομητικό περιεχόμενο. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω το σκεπτικό για την ε, έναρξη ε, μιας πορεία διαπραγματεύσεων για Συμφωνία Ελεύθερων Συλλαγών. Υπάρχουν διάφορα φιλόδοξα διερευνητικά κείμενα τα οποία συμφωνήθηκα την Άνοιξη, τα δώσαμε στην Ίντα, τα στείλαμε στην Επιτροπή Παρακολούθησης τον περασμένο μήνα. Είναι αρκετά λεπτομερή και θα μας επιτρέψουν φυσικά ε, να κάνουμε φιλόδοξες συζητήσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία παρότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες σε τομείς όπως ε, η, ε, τα αγροτικά προϊόντα και οι γεωγραφικές ενδείξεις. Όπως γνωρίζετε η εντολή βρίσκεται στη φάση προετοιμασίας. Πρόκειται για τη σύσταση της ε, απόφασης του Συμβουλίου για, που θα επιτρέψει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις δύο χώρες. Έχουμε το μεταξύ την γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Σιγκαπούρη που βοηθά ε, για το θέμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη. Αυτό βοηθά εμάς και τους εμπορικούς μας εταίρους. Προσβλέπουμε λοιπόν τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των επιπτώσεων αυτής της γνωμοδότησης. Παρά τα θα ολοκληρώσουμε την, την προετοιμασία. Περιμένουμε να υποβάλει η Κομισιόν στο Συμβούλιο σχέδια εντολής μαζί με την έκθεση επιπτώσεων ε, μετά το καλοκαίρι. Θα προχωρήσουμε προς το Συμβούλιο και αφού εγκριθεί από το Συμβούλιο αυτό η εντολή. Θα, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ ήδη από, για την ενθάρρυνσή σας και τις υψηλές σας προσδοκίες. Είναι χώρες που ε, ε, έχουν πάνω κάτω τις ίδιες ιδέες με εμά. Υπάρχουν όρια σε αυτό που σας αντιλαμβάνεστε σε κάποιους τομείς. Αλλά προσβλέπω στη συνεργασία με την ομάδα παρακολούθησης και να σας βοηθήσω εν ώψη της αποστολής σας στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την διπλωματική απάντηση, λέει ο πρόεδρο. ο Ντάνιελ. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, ευχαριστώ πολύ για τις τοποθετήσεις σας. Ε, ζητώ την κατανόησή σας ε, για το ότι δεν κατάφερα να συμπεριλάβω όλες τις προτάσεις σας ε, στο σχέδιο μου. Αλλά θα ήταν και λίγο βαρετό να έχουμε, για παράδειγμα, το κεφάλαιο της βιωσιμότητας και το κεφάλαιο για τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και να μην έχει κανείς να πει τίποτα γι' αυτό. Γιατί τα έχουμε προσθέσει όλα. Εύχομαι να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία τόσο με την Αυστραλία όσο και με τη Νέα Ζηλανδία που να μπορέσουμε να δεχτούμε και να υπερψηφίσουμε. Και αυτή η συζήτηση νομίζω πρέπει να γίνει με κάθε έναν ε, βουλευτή. Δεν γίνεται να υπάρχει εθνικό να, να χρειαστεί να επικυρωθεί η συμφωνία από κάθε εθνικό κοινοβούλιο, από... Δεν ε, πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να κάνουν όλες ε, τις ε, διαδικασίες. Ε. Δεν χρειάζεται να περάσουν οι συμφωνίες αυτές από όλα τα εθνικά κοινοβούλια, έτσι, ώστε να μπορέσουν να τεθούν σε ισχύ. Εμείς είμαστε οι ελεύθερα και δημοκρατικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών, οι οποίοι έχουμε και την αρμοδιότητα να ε, διεξάγουμε αυτές ε, τις ε, διαπραγματεύσεις. Νομίζω πως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όπως και με τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Ελπίζω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί με σαφήνεια και να ε, μιλήσει για το ποιος είναι αρμόδιος, τα Εθνικά Κοινοβούλια εμείς. Μετά, η Επιτροπή Γεωργίας όντως ε, δήλωσε πως θέλει να υποβάλει μια γνωμοδότηση. Εμείς θα χαρούμε για τη συνεισφορά από όλες τις επιτροπές, εφόσον το επιθυμούν. Αλλά ελπίζω να μην συμβεί αυτό που έχουμε δει πολλές φορές, δηλαδή ότι οι άλλες επιτροπές ε, συνειδητοποιούν πολύ αργά ότι θέλουν να, να συνεισφέρουν και αυτές, υπάρχουν καθυστερήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, για να μην λένε στο τέλος ότι δεν προλαβαίνουν, πρέπει να το διευθετήσουμε τώρα το θέμα. Παρακαλώ λοιπόν να μην έχουμε καθυστερήσεις, ακόμα και αν συμμετέχουν και άλλες επιτροπές. Το άλλο θέμα είναι όντως ένα δίλημα. Αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος, ότι η προγραμματισμένη αποστολή μας είναι για τα τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις με το Συμβούλιο γιατί σίγουρα σε αυτήν την περίπτωση θα ζητούσα να υπάρξει μια παράταση, γιατί δεν είναι δυνατόν, δεν θα είναι μάλλον δυνατόν να καταλήξουμε σε μια απόφαση πριν μάθουμε τι προθέσει έχει το Συμβούλιο. Εδώ και τέσσερα ή πέντε χρόνια ζητάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ολοκληρωθεί μια τέτοια συμφωνία Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να είναι επιτέλους σε θέση να το φέρουν εις πέρας. Θα δούμε λοιπόν ε, για την αποστολή της αντιπροσωπείας στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία είμαι θετικά προσκύμενος, θα το δούμε. Να δούμε όμως τι θα γίνει και με την ε, παράταση, αν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή την παράταση ανάλογα με το τι θα κάνει το Συμβούλιο. Ε, αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας και θα χαρώ να λάβω όλες τις τροπολογίες σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τόση μεγάλη χαρά στο τέλος της συνεδρίασης είναι πάρα πολύ καλή αρχή για τις θερινές μας διακοπές. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ το σημείο 25 και το σημείο 26. Σημείο 27, το αγαπημένο μου. Φτάσαμε στα διάφορα. Δεν έχουμε διάφορα. Τίποτα. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 30 και 31 Αυγούστου στις Βρυξέλλες. Καλές διακοπές λοιπόν, να ξεκουραστείτε και να περάσετε καλά.